Eh, Μπορούμε να αρχίσουμε. Ακόμα και αν λείπει η απαρτία, θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 4. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. Μεταδίδεται συνεδρίαση. Άναψα το μικρόφωνο, έτσι. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε ή δεν μ' ακούτε. Μ' ακούτε τώρα. Να, ε, Λειτουργούν τα συστήματα, έχετε διερμηνία, όλα εντάξει. Είναι κακό να μην καταλαβαίνετε τα Ιταλικά. Αλλά υπάρχει φάρμακο. Η γραμματεία το έλυσε το πρόβλημα λοιπόν. Η μερίσια διάταξη στις 14 ε, του μηνός έχει μοιραστεί. Πρέπει το απόγευμα να ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε την έκθεση της Αντιπροέδρου Λεγκρίπ που αφορά το θέμα της εξυγίανσης διαφόρων ιδρυμάτων, διότι αύριο η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα πρέπει ήδη να εξετάσει την έκθεση Φερέιρα και θα πρέπει η γνωμοδότησή μας να υιοθετηθεί απόψε. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τις τροπολογίες που αφορούν την έκθεση Le Grip. Ίσως μπορούμε να συζητήσουμε και την έκθεση Messerschmitt. Δεν θα είναι εύκολο όμως. Μετά την ψηφοφορία μπορούμε να το συζητήσουμε. Η ψηφοφορία είναι έκθεση Εγκρυπ και Σμιτ Θα πρέπει η ψηφοφορία να γίνει κάποιο το πρωί. Μετά έχουμε δική μου γνωμοδότηση για την ερμηνεία του άθρου 202, παράγραφος 5 του κανονισμού που μπορεί να εγκριθεί αύριο το πρωί. Και αυτό και το σημείο 8, έκθεση Χέφνερ για το άρθρο 136 του κανονισμού. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε το απόγευμα, αν μας μένει χρόνος. Να πω τη συνεδρίαση των συντονιστών που προβλεπόταν σήμερα μετά τις 5.30 θα πρέπει να αναβληθεί για αύριο το πρωί στις 9. Διότι δύο εισηγητές των σημαντικότερων ομάδων δεν μπορούν να είναι παρόντες απόψε, θα μπορούν να είναι εδώ αύριο, η Ταρκόσκη και η Γκουαλτιέρη. Γι' αυτό η συνεδρίαση των συντονιστών μπορεί να λάβει χώρα αύριο από τις 9 μέχρι 9.45 και όχι απόψε. Αυτή είναι η ανακοίνωση που είχα να κάνω. να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αύριο την έκθεση Ταρκόφσκη, ίσως μπορούμε να την ψηφίσουμε. Νομίζω ότι έκανα όλες τις ανακοινώσεις που έπρεπε απόψε μετά την ψηφοφορία αν έχουμε χρόνο και θα έχουμε διότι θα έχουμε συντονιστές θα μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεση Γονζέλ που αφορά την αφορμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, πάμε στις ανακοινώσεις. Να επενθυμίσω κάτι σημαντικό. Αύριο ελπίζω να έχουμε περισσότερους παρισταμένους από ότι τώρα. Θα το επαναλάβω αύριο το πρωί, δεν μπορώ να κατηγορώ τους παρόντες για τους απόντες. Αύριο έχουμε έκτατη συνεδρίαση με εκπροσώπους των εκκλησιών και των θρησκευτικών οργανώσεων και των ε, κοσμικών φιλοσοφικών ενώσεων για την εφαρμογή 17 του άρθρου και ε, την εφαρμογή του άρθρου 17 της Συνθήκης της Αβώνας, ενίσχυση της δημοκρατίας είναι το θέμα, της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και πώς μπορεί να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών θα έχουμε και εισηγητές, προσωπικότητες άκρως επιφανεί, όπως ο καθηγητής Βάιλερ, που έγινε πρόεδρος προσφάτως ε, του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ε, του Ευρωπαϊκού και ο καθηγητής Ντερίς του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Όπως είπα, θέλουμε να προωθήσουμε το διάλογο για το άρθρο 17 της Συνθήκης της Αβώνας. Δίνεται στον Αντιπρόεδρο Σουριάν συγκεκριμένη αρμοδιότητα, εκείνος ζήτησε να συνεργαστούμε σαν Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων, να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση και σας παρακαλώ να είστε παρόντες στην συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της ΤΟΑ διαβίβασε μια, ένα δημοσίευμα για τα αποτέλεσματα των ερευνών που ανέθεσε ΣΤΟΑ όσον αφορά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ε, λοιπόν, η ανακοίνωση έγινε μόνο στην αγγλική γλώσσα, υπάρχει μόνο στα αγγλικά και θα λάβετε ένα αντίγραφο δια της ηλεκτρονικής οδού στο σημείο 2 της συνεδριάσεως μας υπάρχει ένα έγγραφο που ετοίμασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν το καθεστώς των κυρώσεων των συνθήκων όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών της 4 Σεπτεμβρίου 2013, 16-17 Σεπτεμβρίου 2013, 14 Οκτωβρίου 2013. Είναι στη διάθεσή σας. Και θεωρούμε ότι εγκρίνονται, διότι δεν έκανε κάποιος κάποια παρατήρηση. Περνάμε αμέσως λοιπόν στην γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου Κωστός Λεγκρίπ αφορά το σημαντικό αυτό ζήτημα της εξυγίανσης των πιστοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων στα πλαίσια ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης και ενός ενιαίου ταμείου εξυγίανσης τραπεζών. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η ΕΚΟΝ έχει την αρμοδιότητα, αύριο πρέπει να αποφασίσει, αλλά η συγγήτριά μας, η κυρία Λεγκρίπ, μπορεί να μιλήσει για την γνωμοδότηση και αναφερθεί στις πολλές τροπολογίες που υπευλήθησαν. 29 τροπολογίες υπευλήθησαν από τους συναδέλφους Νταφ Σούλτς και από την ίδια την κυρία ε, Λεγκρίπ. Της δίνω αμέσω λοιπόν το λόγο. Η κυρία Λεγκρίπ, η συγκήτρια, έχει το λόγο. Σας κατευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημερίζω και τους υπόλοιπους. Σήμερα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για το θέμα της δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης με βάση την Ευρωζώνη. Και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, είναι ζωτικό το θέμα. για την ε, οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας της, πέρα από την Ευρωζώνη, είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού επίλυσης των προβλημάτων ενιαίο. Αυτό είναι ο στόχος της πρότασης κανονισμού που μας προτείνει η Κομισιόν. Είναι κανονισμός που ιδρύει βασικά αυτή την τραπεζική ένωση και αυτή την ενιαία μέθοδο επίλυση εξυγίανσης. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών είναι αρμόδια επί της ουσίας και γι' αυτό θελήσαμε και εμείς εγκαίρως, δηλαδή μέσα στις προβλεπόμενες διορίες, όχι δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο, να γνωμοδοτήσουμε προς την Επιτροπή αυτή. τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης αυτής θα σας τα αναφέρω, έχουν κατατεθεί και ορισμένες τροπολογίες που θα τις αναφέρω συντόμως και αυτές. Τις μελέτησα όλες με μεγάλη προσοχή και ευχαριστώ ένθερμα ιδίως τους κυρίους Νταφ και Σόλτς που έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουν τα πράγματα. Συνολικά λοιπόν Έχουμε 75 τροπολογίες ή 47 για τη γνωμοδότηση και καμιά εικοσαριά από τους συναδέλφους. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι διορίες που υπάρχουν, δεν έχουμε σας είπα πολύ χρόνο, δεν θεώρησα χρήσιμο να οργανώσουμε συνεδρίαση των σκιωδών γιατί επαναλαμβάνω δεν είχαμε πολύ χρόνο. Και απ' την άλλη οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, ορισμένες τουλάχιστον, δεν ήταν προβληματικές αλλά όλες υποστήριζαν και εμπλούτιζαν τις αρχικές ιδέες της ονομαδότησης. Μερικές όμως από τις τροπολογίες αφορούσαν την αύκο καθαρά και γι' αυτό δεν συμβάδιζαν και τόσο πολύ με συμβιβασμούς. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουμε την υποχρέωση να συντάξουμε γνωμοδότηση προς την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή που είναι η αρμόδια επί της ουσίας και πάντοτε θέλαμε εμείς να μην ξεπερνάμε τα όρια των δικαιοδοσιών μας όπως ε, ζητάμε και από τους υπόλοιπους να σέβονται τις αρμοδιότητές μας έτσι θέλουμε να κάνουμε και για τους άλλους. έτσι. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν θέλω να πληροφορήσω την ε, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή χωρίς καθόλου, χωρίς καθόλου να υπερβώ τις δικαιοδοσίες μας. το νέο όργανο ή υπηρεσία, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης δηλαδή, προβλέπει ένα ενιαίο συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, σε με συμμετοχή και εθνικών αρχών και της Κομισιόν. Και αυτό βέβαια θέτει ορισμένα ενδιαφέροντα προβλήματα. που αναφέρονται στο πρώτο, σε ένα από τα τμήματα της πρότασης κανονισμού, το τμήμα 3 που αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Η τίτλοι 1 με 4 του τμήματος 3. Τώρα οι τροπολογίες επικεντρώνονται όλες σε αυτό το τμήμα του κανονισμού. Εγώ φρονώ ε, υποστηρίζω τις τροπολογίες που συγκλίνουν προς ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη λειτουργία αυτή του ενιαίου αυτού διοικητικού συμβουλίου. Υπάρχει πρώτον μία διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου, του διορισμού του Διευθυντή αυτού του Συμβουλίου. Απαιτείται λοιπόν η έγκριση του Κοινοβουλίου και αυτό το λένε οι τροπολογίες 1, 37, 40 και 69 αλλά επίσης 70 και 73 του κυρίου Νταφ και οι 72 του κυρίου Σόλτς προηγούμενες ήταν οι δικές μου. Αυτές όλες μαζί οι τροπολογίες ζητούν περισσότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο για τους διορισμούς για να αυξηθεί έτσι η διαφάνεια και η λογοδοσία, η ευθύνη αυτού του οργάνου. Επίσης υποστηρίζω τις τροπολογίες που ζητούν εγγύηση της εφαρμογής του προγράμματος που θα εγκρίνει το Συμβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν δηλαδή το δικαίωμα να υποβάλουν και αυτά παρατηρήσεις. Είναι οι τροπολογίες 15, 22 και 71 οι δικές μου και οι 67 του κύριου Νταφ. Αυτά πλήρως σύμφωνα με το πρωτόκολλο 1 της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή είναι η δύο κύριοι άξονες των τροπολογιών. Ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω της έγκρισης από το, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποβολή πληροφοριών από και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια. <clears throat> Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο τμήμα τροπολογιών του κυρίου Σόλτς που δεν τις εγκρίνω. Γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο λόγω της σημασίας του θέματος να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, επικεντρωμένοι στις δικές μας δικαιοδοσίες για να πείσουμε έτσι ευκολότερα την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή και την Κομισιόν. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν υποστηρίζω τις τροπολογίες που δεν αναφέρονται άμεσα σε αυτό το θέμα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης αυτού του μελλοντικού ενιαίου μηχανισμού επίλυσης ή εξυγίανσης. Αυτές λοιπόν τις τροπολογίες τις βρίσκω ή υπερβολικά γενικές ή επαναλαμβανόμενες. Και τέλος, με την γνωμοδότηση αυτή αν εγκριθεί, η Επιτροπή μας υπενθυμίζει την στήριξη της για το νομικό υπόβαθρο που προτείνει η Κομισιόν για τον κανονισμό της και το άρθρο 114 της συνθήκης ως υπόβαθρο που προβλέπει την έγκριση μέτρων για την ε, σύγκληση με εθνικά μέτρα. Είναι ε, το άρθρο 114 της συνθήκης που νομίζω ότι, συμφωνεί και γνωμοδότησή μου εξάλλου, ότι είναι η καταλληλότερη νομική βάση με στόχο η διακυβέρνηση αυτή της Τραπεζικής Ένωσης και άρα και του μηχανισμού αυτού με το ταμείο του να συμφωνούν, να συμπεριλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Αυτά είχα να σας πω και θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά σας για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε καταλήλως πληροφορημένοι. Έτσι. μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νταφ ζήτησε να πάρει το λόγο. Τον έχει. Καλό σας απόγευμα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κωνστανση Λεγκρίπ για την παρουσίαση της έκθεσης. Για το θεμελιώδες θέμα της νομικής βάσης ξέρουμε ότι υπάρχει ένα επίμαχο θέμα εδώ, αλλά προς το παρόν το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να επιδείξει σύνεση και να εμείνει στην πρόταση της Κομισιόν και το άρθρο 114 που είναι κατάλληλο και επαρκές για το εγχείρημα αυτό της δημιουργίας του ενιαίου μηχανισμού εξυγένσης. Βέβαια θα αποφασίσει και το δικαστήριο και περιμένουμε να γνωμοδοτήσει. Δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Και τα δύο θα αποφανθούν. Τώρα, κανόνες και διαδικασίες όπως επηρεάζουν εμάς. Για τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ της, των λειτουργιών ενός Εθνικού Κοινοβουλίου από την λειτουργία και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. βέβαια παίζουν ρόλο όταν ε, πρόκειται για τη λογοδοσία των εθνικών αρχών ε, εξυγίανσης και των κυβερνήσεων. Πρέπει να είναι ενήμερα σχετικά με το έργο της ενιαίας αρχής εξυγίανσης, αλλά πρέπει νομίζω να είναι δύο χωριστά τα θέματα αυτά να εδράζονται σε χωριστή βάση από τα θεσμικά ε, όργανα της Ένωσης, γιατί δεν αποτελούν μέρος του νομοθετικού σώματος της Ένωσης. Για να γίνει η διάκριση, κατέθεσα λοιπόν την τροπολογία 67. Τώρα για τη διαδικασία διορισμών Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και το βλέπω και στον κατάλογο ψηφοφοριών στις ε, τροπολογίες 71 και 72 που λέει ότι είναι ταυτόσιμες ενώ όμως δεν είναι και ο κύριος Σόλτσε και εγώ μιλάμε για την ε, σύμφωνη γνώμη ε, ενώ η συγγήτρια μιλάει για έγκριση approval. Μου φαίνεται ότι έχει δίκιο εκείνη και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διατύπωση του κανόνα 109 του εσωτερικού κανονισμού μας που αφορούν το εκτελεστικό συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλλον τίνω λοιπόν να συμφωνήσω με την κυρία Λεγκρίπ και όχι με τη δικιά μου την τροπολογία αν γίνομαι σαφής. Επίσης είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε την ίδια διαδικασία και για τις απολύσεις όπως και για τους διορισμούς και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. για το άρθρο 53, παράγραφος 2, που αφορά το διευθυντή που δεν πρέπει να επηρεάζεται από κανέναν άλλον μου φαίνεται αυτό είναι παράλογο κυρίως διότι στο άρθρο 43 βλέπουμε ότι δεν πρέπει να παίρνει οδηγίες από κανέναν άλλον. Το να λέμε ότι κανείς άλλος δεν θα πρέπει να επιδιώξει να επηρεάσει τον διευθυντή είναι τρελό. συμβουλές θα μπορεί να παίρνει από ενημερωμένες και έγκυρες πηγές. Καλό είναι λοιπόν να διαγράψουμε την παράγραφο 2 του άρθρου 53. Και στο τέλος, ε, στην τροπολογία 75, προσπαθώ να προσθέσω μία παράγραφο που θα προβλέπει μία διαδικασία επανεξέτασης του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης για να μπορεί ο μηχανισμός ε, εξυγίανσης να λειτουργεί σαν μέσον προστασίας και θωράκισης για τις τράπεζες, γιατί κάνουμε λάθος αν θεωρούμε ότι οι εθνικές αρχές εξυγίανσης και οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την εξουσία να μπλοκάρουν τις αποφάσεις του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης σχετικά με το κλείσιμο και την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Ο ενιαίος μηχανισμός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας υπάρχει και θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Ε, δεν νομίζω γιατί ε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο ε, να δημιουργηθεί για την κρίση των τραπεζών και την αντιμετώπιση της πέρα από τον ESM. Καλό είναι να υπάρχει όμως και στον κανονισμό πρόβλεψη για διαδικασία ε, πανεξέτασης ή αναθεώρησης. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε την έννοια της επανεξέτασης και να της δώσουμε και την κατεύθυνση που θέλουμε. Ευχαριστώ κύριε Ντόφ. Ο μπρονξ είναι επόμενος που θα πάρει το λόγο. Ο κ. Μπρόνξ. Τα σχόλιά μου απευθύνονται πιο πολύ προς εκείνους στη χώρα μου που περνούν τόσο ήσυχη ζωή που ξαδεύουν το απόγευμα τους παρατηρώντας εμάς, παρακολουθώντας εμάς και όχι στους ευρωβουλευτές που είναι παρόντες, διότι οι πρώτοι είναι πιο πολύ άριθμοι από τους δεύτερους. Υπάρχουν κάποιοι στη χώρα μου που ίσως διερωτώνται γιατί συμμετέχω σε αδίποτε συζήτηση, γιατί ψηφίζω, διότι επηρεάζει μόνο χώρε τη Ευρωζώνη. οι άλλε συμμετέχουσε χώρε και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι στην Ευρωζώνη και είναι απίθανο να συμμετάσχει και σαν χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μελλοντική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα σε στο στόχο την είσοδο στην Ευρωζώνη ή να συμμετέχει σαν χώρα. Λοιπόν, και ο κανόνες για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η εξαίρεση μη συμμετοχών των κρατών μελών δεν ισχύει για το Κοινοβούλιο. Άρα έχω δικαίωμα να συμμετέχω και καθήκον ίσω, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Θέλουμε να προωθήσουμε και να επεσπιστούμε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων αλλά δεν ξεκινά, δεν περιορίζεται στο ρόλο του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να υπερασπιστώ και να προωθήσω το ρόλο εθνικών κοινοβουλίων όλων των κάτων μελών. Λοιπόν, δεν, είμαι, δεν περιορίζομαι τόσο στα Βρετανικά. Είμαι ενθουσιώδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλω να παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπερψηφίσω τι τροπολογίε που αυξάνουν το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα καταψηφίσω τι τροπολογίε που μειώνουν το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είμαι ενθουσιώδη υποστηριξή του, του Συμβουλίου, αλλά τουλάχιστον συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών. Λιγότερο ενθουσιώδη είμαι για το Κοινοβούλιο όταν ασκεί εξουσίε επί των κρατών μελών. Όμως είμαι υπέρ του Κοινοβουλίου διότι είναι εκλεγμένο σώμα και ελέγχει διορισμένους φορείς όπως ε, ο προτινόμενο, το προτινόμενο Διοικητικό Συμβουλίο του Μηχανισμού ε, Εξυγίανσης. Αλλιώς θα ήταν ανεξέλεγκτος αυτός ο φορέας. Γι' αυτό θα υποψηφίσω τις σχετικές τροπολογίες που αυξάνουν τον έλεγχο. Θα απόσχω από υποβολή άλλων ε, τροπολογίες που αφορούν το κείμενο, τη σύνταξη, και εκτιμώ και τις άλλες απόψεις και τις απόψεις των άλλων κατών μελών και όχι μόνο της δικής μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μορέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντική έκθεση αυτή. Είναι από τις πιο αποφασιστικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες της κρίσης. Ε, τραπεζική Ένωση στην Ευρώπη με νέο μηχανισμό εξυγίανσης. Είναι πράγματι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και η γνωμοδότησή μας σχετικά με τη συνταγματική πλευρά της πρωτοβουλίας αυτής θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ σημαντική συνεισφορά στον κανονισμό. Ε, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να διευκρινίσει το συνταγματικό το θεσμικό καθεστώς ε, του ενιαίου μηχανισμού. αρχίζοντα από τη νομική βάση, δεν είμαι βέβαιος ότι η βάση αυτή είναι επαρκής. Γιατί το 114 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στην προσέγγιση της εθνικής νομοθεσίας αναφερόμενοι στην δημιουργία και λειτουργία της ενίας αγοράς. Και αναρωτιέμαι αν η θέσπιση καινούριου νέου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου θα μπορούσε να καλύπτεται από αυτή τη νομική βάση. Αλλά φοβούμαι ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε ευρέως εκτατικά το άρθρο αυτό σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας περιμένουμε τι θα πει και το δικαστήριο. Δεν είμαι βέβαιος αν θα θεωρήσει το δικαστήριο επαρκή αυτή τη νομική βάση. Ίσως εδώ είναι μια περίπτωση όπου χρειάζεται αναθεώρηση της συνθήκης κατεπηγόντως για να προσθέσουμε όχι μόνο αυτά που κάνουμε στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης και την ε, ρύθμιση ε, χρηματοπιστωτικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για να επιτρέπουμε να λαμβάνονται και περισσότερες αποφάσεις για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του ρόλου του δικού μας Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Η εκτελεστική ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να είναι υπόλογη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι ενώπιον των εθνικών. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν μπορεί να είναι υπόλογα μπροστά στα εθνικά κοινοβούλια. Τα τελευταία έχουν το δικό τους ρόλο βάσει της συνθήκης ε, και κυρίως της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται. Οι προτάσεις τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αλλά ένα είναι αυτό και άλλο είναι το θέμα της λογοδοσίας που σημαίνει ότι ένα σώμα είναι υπεύθυνο και λογοδοτεί μπροστά σε ένα κοινοβούλιο. Αυτό δεν ισχύει για τα εθνικά κοινοβούλια. Θέλω λοιπόν σαφή διάκριση μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους διορισμούς και τις απολύσεις των ε, μελών του SRM, του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγένσης, πιστεύω και εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία και ο ρόλος του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι ο ίδιος σχετικά με προσλήψεις και απολύσεις και πιο σωστό είναι να μιλήσουμε για έγκριση approval παρά για σύμφωνη γνώμη συγκατάθεση consent. όχι να συγκατατίθεται στο Συμβούλιο, αλλά να συμμερίζεται τις αποφάσεις για ε, διορισμούς και απολύσεις. Οπότε και εδώ συμφωνώ με τις απόψεις του συναδέλφου Νταφ. Και τέλος, είναι εξαιρετικό το έργο της εισηγήτριας και το, το, καλό έργο πρέπει να το επενούμε. Γι' αυτό γενικά στηρίζουμε την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Η συγκήτρια ίσως θέλει να ασκήσει το δικαίωμά της να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν. Η κυρία Λεγκρίπ λοιπόν έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους τρεις συναδέλφους που Φράστηκαν για την γενική τους υποστήριξη στο σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν και ο κύριος Μορέιρα και ο κύριος Νταφ. Βέβαια όντως χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς την οικοδόμηση της, Ευρωπαϊ... της Τραπεζικής Ένωσης. αν εγκριθεί αυτή η γνωμοδότηση συμβάλλουμε και εμείς λιγάκι στον δρόμο αυτόν που θα είναι μακρύς. Τώρα αρχίζει απλώς η διαδικασία. Καλώς. Ε, κλείνει η συζήτηση. Α, ο κύριος Νταφ θέλει να πει κάτι. Έχετε το λόγο. Α. Ναι. Ζητώ συγγνώμη που δεύτερο λόγο. για τη νομική βάση θέλω να πω τη νομική βάση της πρότασης η γερμανική κυβέρνηση από ό,τι γνωρίζω ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 352 το 114 αντικαταστήσουμε το 352 η δική μου άποψη είναι εξή. όπως υπονόησε ο κύριος Μορέιρα θεωρώ ότι αν προχωρήσουμε με τον κανονισμό υπ' αυτή τη μορφή, αυτό είναι πρώτο βήμα απλώς. Ένα πρώτο βήμα προς ομοσπονδιακό μηχανισμό εξυγίανσης όπως θα μπορούσε να αποκληθεί. Εν ευθέτω χρόνο και πιο καλά σύντομα Ίσως θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση της συνθήκης για να καλυφθεί και να ρυθμιστεί αυτή η προσέγγιση. Η ίδρυση ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης αφορά μεγάλη μεταφορά κυριαρχίας από τα κράτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτή την κίνηση να τη συμπιέσουμε στους περιορισμούς της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ταχύ σαν προσέγγιση που αρμόζει σε προσωρινό μέτρο αλλά δεν είναι κάτι βιώσιμο σαν βάση για κάτι τόσο σημαντικό για μια τόσο μεγάλη εμβάθυνση και ε, όσον αφορά την οικονομική ολοκλήρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξαναπάτε το λόγο κυρία Λεγκρίπ. Δεν απομένει παρά να περιμένουμε τέσσερα λεπτά σύμφωνα με το ρολόι μου για να πάμε στην ψηφοφορία ελπίζοντας να καταφτάσουν εντωμεταξύ και άλλοι συνάδελφοι. Διακόπτουμε λοιπόν για ένα πεντάλεπτο. I... Πρόεδρε, μήπως μπορούμε να προχωρήσουμε. In effetti possiamo cominciare come chiede Μπορούμε να ξεκινήσουμε, όπως έλεγε και ο συνάδελφος Νταφ, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την εξυγίανση των χρηματοστικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο του ενίου μηχανισμού εξυγίανσης ενός ενιαίου ταμείου εξυγίανσης τράπεζων που τροποποιεί τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Λοιπόν, ψηφίζουμε Τροπολογία 58. Σόλτς. Υπέρ. Σήκωσα το χέρι. Κατά. Απορρίπτεται. Ορίστε. Ψηφίσαμε, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 58. Ψηφίστηκε. Θέλετε να πάρετε τροπολογία την επόμενη. Α, Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Α, δηλώσατε αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν με μια αποχή, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 59, υπέρ. Κατά. Καμία αποχή. Α, μία αποχή. Τροπολογία 60, Σόλτς, υπέρ. Κατά. Αποχές μία αποχή. Τροπολογία 61, Σόλτς, υπέρ. Κατά, άποχες, μία αποχή. 62, Σόλτς, υπέρ. Κατά, αποχές, μία υπέρ. Πρόεδρε, ορίστε. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Αν μπορείτε να μας λέτε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σε κάθε περίπτωση, διότι δεν το κάνετε αυτό, δεν μας λέτε αν απορρίπτεται, εγκρίνεται κάθε τροπολογία. Α, ναι. Μου υπενθυμίζετε ένα καθήκον. Είναι προφανές βέβαια. Λοιπόν, όλες οι τροπολογίες μέχρι τώρα, Σόλτς, έχουν απορριφθεί εκτός από μία περίπτωση. Όλες απερίφθησαν με αποχή εκτός από μία ψήφο θετική που είχαμε. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά μία εποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 9, 10, 11, 12 είναι προφορική. Αφορούν διορθώσεις του κειμένου και δεν ψηφίζονται. Τροπολογία 13 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της ηγήτριας υπέρ. κατά άποχες εγκρίνεται 65 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 16 της ηγήτριας υπέρ κατά να επαναλάβουμε. Δεν είναι ξεκαθάρο. Τροπολογία 16 της ηγήτριας, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 και 18 μπορούν να ψηφιστούν μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 67 και τα δύο τμήματα καταπίπτουν, δεν ψηφίζουμε την 67. Πάμε στη 19, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 διορθωτική του κειμένου δεν ψηφίζουμε τροπολογία 21 συμπληρωματική 25 ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Είπε κανείς κάτι. Και δύο τροπολογίες και 21 και 25 εγκρίθηκαν. 25 λέει ο πρόεδρος, ψηφίστηκε μαζί. Εγκρίνεται και 25, ναι, ναι, ναι. 22 τσιγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 και 24 αφορούν το κείμενο, κάνουν διορθώσεις, άρα δεν ψηφίζονται. Την 25 ήδη εγκρίθηκε μαζί με την 21, 26 υπέρ. Μετά, αποχές εγκρίνεται. 27 αφορά διορθώσεις και αυτή. Δεν ψηφίζουμε. Τοπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 ψηφίζουμε την 29 στην πράξη ψηφίζουμε μαζί και την 33 και την 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνονται λοιπόν 29, 33 και 37 Τροπολογία 30 και 31 και 32 διόρθων το κείμενο, άρα δεν ψηφίζουμε. 33 ήδη ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στην ομάδα. 34 ψηφίζουμε υπέρ. Κάτα. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 35 διότι αφορά διόρθωση του κειμένου. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 και αυτή ψηφίστηκε στην ομάδα των τροπολογιών εγκρίνεται λοιπόν 68 καταπίπτει διότι εγκρίθηκε 37 38 διορθώνει το κείμενο δεν ψηφίζουμε 69 Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. κατέπεσε 70 διότι εγκρίθηκε η 71 και 72 είναι ταυτόσιμες ήδη εγκρίθηκα άρα καταπίπτει η 70 ορίστε λυπάμαι λέει ο κ. Ντόφ όπως εξήγησα όταν πήρα το λόγο δεν είναι ταυτόσιμες περάσαμε όμως την 71 Πιθανότατα οι 72 και οι 70 και οι 39 τώρα είναι, έχουν καταπέσει. Πάμε στη 41 τώρα, συνεπώς. Σας ευχαριστώ. Είπα ότι δεν είναι με 72 και καταπίπτει. Συμφωνούμε. Ψηφίζουμε την 41 διότι 40 φορά διόρθωση και δεν ψηφίζεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι γίνεται. αυτό τη γραμματεία. 73-42 για μένα λέει ότι 42 καταπίπτει 73 εγκρίνεται. Κατά άποψή μου, διάβασα την 73 και 42 και θεωρώ ότι είναι ταυτόσιμε οι τροπολογίε Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα να καταπέσει η 42. 43, 42 συγγνώμη και 73 θεωρώ ότι είναι ταυτόσιμες λέει ο πρόεδρος. Comunque non cambia la sostanza, eh? Δεν αλλάζει η ουσία όμως για να μην χρονοτριβούμε. Ψηφίζουμε την 73. Ο Νταφ, κύριος Νταφ, πρόεδρε. Θα, Θα ήθελα να αποσύρω την 73. Α, εντάξει. Λοιπόν, αποσύρεται 73 και ψηφίζουμε μόνο τη 42. Υπέρ, σηκώστε το χέρι παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 74. Ταφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές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 Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54. Σόλτς υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 λεγκρίπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 λεγκρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν 15 υπέρ μία εναντίον και καμία αποχή ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Λεγκρίπ για τη δουλειά της ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης Δεν βλέπω όμως τον συνάδελφο Μέσο Σμιτ. Παρακαλώ λοιπόν τον συνάδελφο Ραντζέλ να δεχτεί να συζητήσουμε τώρα την έκθεση τη σχετική όσον αφορά την επικαιροποίηση της συνθήκης της Αβώνας. Ε, εξυγχρονισμό όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κανονικά θα συζητούσαμε το θέμα αύριο. Αλλά και στην αρχή της συνεδρίασης είπα ότι μπορεί να μετακινηθεί και να συζητηθεί το απόγευμα, αν έχουμε χρόνο. Και εφόσον βρίσκεται ο συνάδελφος Ράντζελ που έχει μελετήσει το θέμα, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα α, ε, για δημόσια κρόση που θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου του 2014 για το θέμα αυτό. Οπότε μπορεί να μας ενημερώσει ο συνάδελφος Ραντζέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Εκτός προγράμματος. Για να μιλήσω αγγλικά θα πρέπει να έχω χρόνο να προετοιμαστώ. Ε, στα πορτογαλικά λοιπόν. Κάνα μισά ώρα σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά προετοιμαστεί. Όπως ξέρουν όλοι λοιπόν, αυτό που εμέσως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των συντονιστών των πολιτικών ομάδων ήταν ότι αυτή η έκθεση η οποία αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας δεν μπαίνει σε όλα τα θέματα που καλύπτονται από αυτό το πλαίσιο, ούτε μιλάει για τα, το διοργανικό πλαίσιο μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Αυτό που αποφασίσαμε, και αυτή ήταν συμφωνία μεταξύ όλων, συμφωνήσαμε λοιπόν ο κύριος Λαμασούρ να αναλάβει τη σχέση με το Συμβούλιο γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα και με μια πιο γενική έννοια η έκθεση Τσαρσκόφσκι Γκουαλτιέρη αφορά τα πολυεπίπεδα θέματα, πολλαπλά επίπεδα, διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης δηλαδή ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μπορεί αργότερα να γίνει και έκθεση για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ πάντως τώρα θα πιάσω την συνθήκη της Λισαβόνας και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί. Αυτά συμφωνήσαμε. Ε, βέβαια μπορεί να υπάρξουν αλλαγές αργότερα αν αποφασίσουμε να κάνουμε αλλαγές. Αλλά γενικά εγώ θα επικεντρωθώ στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο που σημειώνουμε είναι ότι στην επιστολή για τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν αναφέρονται φιλόδοξα πράγματα σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το Κοινοβούλιο σαφέστατα κέρδισε ε, πολιτικές, θεσμικές, συνταγματικές εξουσίες μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας εξουσίες που το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ασκεί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και, και, άλλες που δεν τις είχε πριν. Αν λοιπόν το δούμε μαξιμαλιστικά, βλέπουμε ότι βελτιώνονται πολύ οι, εξωτε... οι εξουσίες του Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι το Συμβούλιο προσπαθούσε να μεγιστοποιήσει τη δική του τη θέση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιζε ρόλο ενδιάμεσου, μεσάζοντα. Και το Κοινοβούλιο βρέθηκε ε, σφινωμένο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τάσεις. Δηλαδή ο ρόλος του μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας και η προσπάθεια του Συμβουλίου για διαφορετική ερμηνεία. Και αυτό είναι ο ρόλος που βλέπει τώρα ε, να έχει το, το Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι η πολιτική βάση της έκθεσής μου. Για να δούμε τώρα τη, τα καινοφανή από την Κομισιόν. Ο πρόεδρος της Κομισιόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκλέγει, όχι πια να εγκρίνει, αλλά να εκλέγει τον υποψήφιο. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Ε, υπήρχε δυνατότητα να καταργείται η Κομισιόν. Από το 1979 ε, υπήρξαν και εγκρίθηκαν πολλές εκθέσεις που έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια ότι η Κομισιόν ε, ενίσχυσε το ρόλο και βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία της, θα πρέπει να υπάρχει μια αντιρρόπηση. Και στην πορεία των ετών έγιναν διάφορα δημοψηφίσματα, εκείνο της Ιρλανδίας για παράδειγμα, που αποφάσισε να αλλάξει τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ώστε και γεωπολιτικά να υπάρχει ε, μια ε, αντανάκλαση των συσχετισμών στην Κομισιόν, αλλά το Συμβούλιο αρνήθηκε και προσπάθησαν να βρουν μια μέση λύση και να ικανοποιήσουν τους Ιρλανδούς και να δημιουργήσουν αυτό το σχέδιο ad hoc που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το ιστορικό. Υπήρξαν δύο βασικές αλλαγές σημαντικές στη λειτουργία της Κομισιόν. Τώρα, είναι σαφές ότι η Κομισιόν έχει χάσει λίγο έδαφος. Αυτό είναι κακό από την άποψη της ε, Ομοσπονδίας ή της ολοκλήρωσης. Δεν εξυπηρετεί δηλαδή αυτά. Αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, φαίνεται αυτό. Αυτό που πρέπει να αναλύσουμε όμως σε αυτό το στάδιο είναι πώς η Κομισιόν διορίζεται, ορίζεται ή πώς γίνεται η σύνθεσή της. Μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζωτικό ρόλο σε σχέση στα πλαίσια τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο ρόλος μας είναι κέριο και γι' αυτό πρέπει να δούμε πολλές λεπτομέρειες και τώρα μέχρι τι εκλογέ. και θα πρέπει μετά το Μάιο-Ιούνιο να τεστάρουμε το καινούριο σύστημα. Οπότε ε, έχουμε ένα βασικό τεστ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις καινούριες εξουσίες. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή το ειδικό βάρος αυτό του Κοινοβουλίου ποιο ακριβώς είναι. Και νομίζω ότι ο, ένας απολογισμός είναι θετικός. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αρχίζουν να προτείνουν υποψηφίους για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις εκλογές. Ξέρουμε ότι έχουμε το ψήφισμα του 2012 του Κοινοβουλίου που έλεγε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εκλέγονται μέσα από ένα πλαίσιο που θα εδράζεται σε δημοκρατικές αρχές. Και αυτό πάλι ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν προταθούν πριν από τις εκλογές στα μέλη της Επιτροπής, υπάρχει μεγαλύτερη, αν γίνεται από πριν η εκλογή, υπάρχει περιθώριο ελιγμών και ενισχύεται η δημοκρατική διαδικασία. Έμεσα όμως μέσα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίση μπορεί με αυτό το σύστημα τα πιθανά μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν τρόπον την στις ευρωπαϊκές εκλογές και να ψηφίζονται. Να... Και αυτό είναι πολύ θετικό δηλαδή να παλεύουν, να δίνουν μάχη για την ψήφο των πολιτών. Είναι καλό αυτό, αν και είναι μια παράλληλη λογική προς ε, τη δική μας θεσμική και συνταγματική ε, μορφή. Μπορεί λοιπόν να είναι μέτρα παρασυνταγματικά αυτά που λαμβάνονται για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και νομιμοποίηση. Μια και μιλάμε για τη δημοκρατική νομιμότητα για την Κομισιόν, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μπορεί αυτή να ενισχυθεί ακόμα περισσότερα. δεν ξέρω πώς ακριβώς. Αλλά είναι ένας λόγος για να το συζητήσουμε. Πολλοί σκέφτονται να μειώσουν το βάρος και τη σημασία της Κομισιόν. Αν όμως πρόκειται να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν ή ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ε, για να έχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα τεθεί προς αναθεώρηση η συνθήκη. Με δεδομένο τις συνθήκες που έχουμε και με δεδομένο αυτά που ακούσαμε στους διαδρόμους και στα παρασκήνια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων υπάρχουν πιθανές κινήσεις προς τα μπρος και καλό είναι να, αρχίζουμε, να αρχίσουμε από τώρα να προλυαίνουμε το έδαφος γι' αυτό. Έχουμε ε, ορισμένες θετικές αλλαγές που προτείνονται για να θα ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό ρόλο στην ε, ε, εκλογή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την Κομισιόν. Αυτό είναι ένα βήμα. Να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό βέβαια μια ενδιαφέρουσα πρόταση που χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας είναι για παράδειγμα η εξής. να απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου για να γίνει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν απαιτείται μόνο πλειοψηφία με ένα καινούριο σύστημα, αλλά απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Η αλλαγή του συστήματος διασφαλίζει ότι μια απλή πλειοψηφία μπορεί να επιφέρει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κομμάτι της πολυεπίπεδης προσέγγισης που εξετάζει διάφορες αλληλεπιδράσεις και αλληλένδετες σχέσεις στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Αυτό είναι σημαντικό. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να ε, εκφράζει ψήφο δυσπιστίας ή μη εμπιστοσύνη ε, σε έναν επίτροπο. Έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ε, καταργεί, να καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήμουν κατά των μεμονωμένων ψήφων μη εμπιστοσύνης. Γιατί? Γιατί αντιτάσσεται στην εμπειρία που είχαμε από τη Συμφωνία Πλαίσιο και όλες τις διαπραγματεύσεις μας. Αυτό πρέπει να το ε, αναγνωρίσουμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια φορά την αδυναμία του Κοινοβουλίου. Καμιά φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια πολύ μετριοπαθή αντίληψη σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών. Λέμε πολλές φορές ότι θα έπρεπε να συνοδεύουμε τους διεθνείς ε, διαπραγματευτές, σαν να είμαστε εμείς διεθνείς διαπραγματευτές. Δεν υπάρχει διεθνές πρόγραμμα ή σχέδιο που τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου παρακολουθούν σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να δώσουν την έγκρισή τους ή όχι μετά από ψήφο ή κάποιο είδους δημοψήφισμα, αλλά δεν παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις. Δεν βοηθάει αυτό. Βέβαια μπορεί εδώ να είμαι η μειοψηφία. Λένε όλοι ότι πρέπει να συμμετέχουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι παράδοξο, γιατί πουθενά δεν πάνε οι βουλευτές ε, οι ίδιοι να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια μικρή ομάδα στα πλαίσια μιας εντολής που έδωσε το Κοινοβούλιο, αλλά δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Μετέχουν μέσα από τη διαδικασία της επικύρωσης. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα έχουμε μπερδεμένα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα ε, να αποφασίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς ποιος είναι και ποιος δεν είναι ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μιας κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα προνόμιο που θα πρέπει να ασκείται από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ε, καθίσουμε εμείς εδώ και πούμε ότι να έχουμε ας πούμε μια κυβέρνηση η οποία θα καθοδηγείται από τη συνέλευση, ε, δηλαδή για να αποφύγουμε την τρομοκρατία μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αν έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση ε, που θα διέπεται από τη και θα κυβερνάται από τη συνέλευση, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν θα υπάρχει η αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας. Αν αποφασίζει το κοινοβούλιο ποιος θα μετέχει και ποιος δεν θα μετέχει στην κυβέρνηση με καζουιστικό τρόπο, τότε ε, δεν θα μπορούμε να πούμε τι ε, Ακριβώ θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρόκειται για κυβέρνηση που θα καθοδηγείται από τη συνέλευση, από το Κοινοβούλιο. Εδώ το πιο χαρακτηριστικό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει μια κυβέρνηση ε, που επηρεάζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ε, και υπάρχει και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέλο πάντων, ε, δεν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εμεί έχουμε αναλογική εκπροσώπηση και όχι πλειοψηφικό όπω το Ηνωμένο Βασίλειο τρόπον την είναι κατακαιρματισμένη η προσέγγιση μας. Εγώ πάντως με αυτό το παράδειγμα ήθελα να δείξω ότι, αυτή ότι πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση υπονομεύει και κατακαιρματίζει την εκτελεστική εξουσία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε δημοκρατικό έλεγχο στην Κομισιόν. Και αυτό είναι ο κανόνας της απόλυτης πλειοψηφίας για την ε, κατάργηση της ε, Επιτροπής είναι καλός δεν επηρεάζομαι την καθημερινή δουλειά της ε, Κομισιόν. Το να έχουμε ε, τη δυνατότητα ψήφου μη εμπιστοσύνη ε, απέναντι σε μέλη της Επιτροπής, σε μεμονωμένους επιτρόπους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική παρέμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξωτερικές διαπραγματεύσεις της Κομισιόν. Άλλο είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο και άλλο είναι να πάμε να αυθαίρετα να διώχνουμε μέλη τη Επιτροπή. Θα ήθελα να καταδείξω ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζομαι τώρα. Ένα πρόβλημα όπου τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων παρεμβαίνουν ε, σε διαπραγματεύσεις ευρωπαϊκές και διεθνείς. Η Άγγελα Μέρκελ, για παράδειγμα, θέλει να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, να πάει στο, στο κοινοβούλιο της και να συζητήσει. Και αυτό καθυστερεί τη διαδικασία. Και έχουμε την εντύπωση στην Ευρώπη ότι οι κυβερνήσεις ελέγχονται απόλυτα από τα εθνικά κοινοβούλια ή τις εθνοσυνελεύσεις τους. Και κανείς δεν κερδίζει όταν έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει και αυτή ε, στην ιδιωτική της σφαίρα της εξουσίας της χωρίς πολλές ε, ξένες παρεμβάσεις Πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών. Εξετάζομαι λοιπόν τις εξουσίες Κοινοβουλίου και Κομισιόν για να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και ίσως μπορούμε τις νομοθετικές εξουσίες και τις πρωτοβουλίες για ανάληψη νομοθετικών προτάσεων να τις ενισχύσουμε και αυτές. Δεν θέλουμε όμως να ε, αποφασίζει ε, για, και, να καθοδηγεί την κυβέρνηση το Κοινοβούλιο και τα μέλη του. Επίσης, επειδή μιλάμε και για την αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας, πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που εγκαταλείψαμε ε, στη συνταγματική συνθήκη, δηλαδή ε, το πώς ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγει, επιλέγει τους επιτρόπους. Καλό θα ήταν να επαναφέρουμε ίσως την ιδέα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ζητάει κάθε κράτος μέλος να του ορίσουν τρεις και να διαλέξει ο πρόεδρος ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις. Γιατί πρώτος, πρώτον και πρώτιστα θα υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλονται και τα δύο φύλλα, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων το θέλουμε αυτό πολύ. Θα είναι πλουραλιστές και θα διαλέγουν υποψήφιους και από τα δύο φύλλα. Και έτσι θα λυθεί αυτό κατευθείαν. Επίσης θα γίνεται καλύτερο συντονισμός των χαρτοφυλακίων. Φανταστείτε μια περίπτωση όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, ε, δίδει, αναθέτει τα χαρτοφυλάκια με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα των προτινομένων. Είναι δύσκολο ο πρόεδρος της Επιτροπής να αναθέσει χαρτοφυλάκια άμα δεν ξέρει τα ε, προσόντα. Άρα θα βελτιωθεί έτσι ο συντονισμός της διαδικασίας ανάθεσης των χαρτοφυλακίων. Ε, μια οδός που είναι λίγο επικίνδυνη είναι να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική προσέγγιση. Τι δηλαδή. Να ενισχύσουμε την ικανότητα, την πολιτική ικανότητα των ευρωπαϊκών κομμάτων να ορίζουν υποψηφίους για προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, προσεγγίσουμε το βρετανικό ας πούμε μοντέλο όπου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προέρχονται από το Κοινοβούλιο. Θα έχουν εκλεγεί από αυτό το σώμα για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ε, εγώ δεν θα ήθελα να ψηφίζομαι μεμονωμένα ε, και να δίνομαι ψήφο μη εμπιστοσύνη, γιατί έτσι παρεμβαίνουμε υπέρμετρα στο έργο της Κομισιόν. Όμως θα έδινα στον πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την επιλογή να διαλέξει μεταξύ τριών προτινομένων από το κράτος μέλος. Και μετά μπορούμε να θεσπίσουμε ένα κανόνα ε, όπου, που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να δίνει ψήφο μη εμπιστοσύνη ε, με όχι απλή πλειοψηφία όμως, αλλά πλειοψηφία των δύο τρίτων για λόγους με καλύτερη σταθερότητα. Δηλαδή θα, προσ... θα, θα δεν θα χορηγείτε δηλαδή, δεν θα δίνεται ψήφος ε, μη εμπιστοσύνη, αλλά θα μπορεί το Κοινοβούλιο να ανατρέψει ή να ε, ζητήσει να προσαχθεί στην ε, δικαιοσύνη μέλος της Επιτροπής. Συγκρίνω εδώ δηλαδή το βρετανικό μοντέλο και το αμερικανικό. Αν δούμε το βρετανικό, της 17ου και 18ου αιώνα ήταν μοντέλο προσαγωγής αλλά απαιτούσε απλή πλειοψηφία. Δηλαδή το σύστημα έγινε στο τέλος ένα κοινοβουλευτικό μοντέλο. Δηλαδή ε, ε χρησιμοποιήθηκε το ε, κοινοβούλιο για την προσαγωγή. Τα δύο τρίτα στην Αμερική διατηρήθηκαν ε, για την απαγγελία κατηγοριών. Στην Αμερική έγινε πιο προεδρικό το μοντέλο έτσι. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτής της αυξημένης και ενισχυμένης κοινοβουλευτικής προσέγγισης. Πρώτον, εδώ θα δημιουργούσαμε έναν άξονα Επιτροπής Κοινοβουλίου θα είχαμε ένα συνταγματικό συνεχές μεταξύ, κοινοβουλίου και, μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και αυτό θα σήμαινε ότι ο άλλος πόλος της πολιτικής έντασης και ο άλλος πόλος των συνταγματικών εξουσιών θα ήταν το Συμβούλιο. Και αν σήμερα έχουμε ανησυχίες και προβλήματα ε, λόγω δυσαναλογιών και ε, μεγάλων αυξήσεων των εξουσιών του Συμβουλίου μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, Ξέρουμε ότι αυτό οφείλεται σε δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, οφείλεται στην κρίση που δεν είχε προβλεφθεί από τις συνθήκες, κάτι το οποίο τώρα λύνεται με διακυβερνητικές μεθόδους και ένα δεύτερο παράγοντα διαφορετικό, μια μαξιμαλιστική ερμηνεία των συνθήκων από το Συμβούλιο. Αυτό ε, θα μπορούσε να προβλεφθεί από ανθρώπους όπως εγώ, που εξετάζαμε τις συμφωνίες πλαίσιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων και έπρεπε συνεχώς να κάνουμε πίσω και να λέμε όχι δεν ήταν αυτή ε, η, πρόθεση. Ήταν θέμα ερμηνείας. Ε, αν λοιπόν υπάρχει αυτό το μεγάλο μέλημα ότι το Συμβούλιο ε, αύξησε υπερβολικά τις εξουσίες, μπορεί να δούμε ότι τώρα μπαίνει σε μια συνταγματική σύγκρουση το Συμβούλιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν την Ένωση. Ε, και δημιουργείται ε, αυτό το συνεχές μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Κομισιόν και ε, το Κοινοβούλιο εδώ εκπροσωπεί τους λαούς και τις κυβερνήσεις ε, η Κομισιόν. Ε, υπάρχει λοιπόν, δημιουργείται ένα, έτσι, σχίσμα μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Ε, δεν λέω ότι η κοινοβουλευτική προσέγγιση μπορεί να είναι λάθος, αλλά δημιουργεί κάποια σχιζοφρένεια, διότι υπάρχουν τα σώματα που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των κρατών μελών και θα πρέπει να είναι κομμάτι της αρχιτεκτονικής, η αντιπροσώπευση δηλαδή, η εκπροσώπηση των κρατών μελών, που, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έπρεπε να είναι σε ελεύθερη τροχιά αλλά να υπάρχει ε, να υπάρχουν ίσοι κανόνες του παιχνιδιού ε, ό,τι αφορά ε, την λειτουργία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ποια εναλλακτική λύση υπάρχει ή ποιος αντιρροπιστικός μηχανισμός Ξέρουμε ότι η αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας είναι θέμα κλειδί και αυτό προσπάθησα να το αναδείξω εδώ. Αν θέλουμε να έχει αυτονομία η εκτελεστική εξουσία και αν ενδεχομένως θέλουμε να ενισχύσουμε τις εξουσίες της Κομισιόν ε, μαζί με το Συμβούλιο και θέλουμε να αποφύγουμε αυτή την ορατή ε, ε, ε, ε, αυτή τη διαφορά, τη σύγκρουση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σώματα που εκπροσωπούν πολίτες και οργανωμένα ευρωπαϊκά συμφέροντα πολιτών, μπορούμε, αντί να ακολουθήσουμε την κοινοβουλευτική οδό, να ακολουθήσουμε μια πιο προεδρική οδό σε σχέση να, να έχουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος θα θυμίζει περισσότερο προεδρική προσωπικότητα, πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Και είναι σημαντικό, να το πούμε και αυτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, Να σας δώσω μια εικόνα που βοηθάει, νομίζω, γιατί είναι δύσκολο τα μοντέλα αυτά διακυβέρνησης να τα εφαρμόζουμε όταν τα ξέρουμε από τα κράτη-μέλη μας ή από τις ομοσπονδίες μας και να πάμε να τα εφαρμόσουμε σε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, είναι ε, μια σειρά θεσμικών οργάνων και κάθε θεσμικό όργανο έχει ε, μια μοναδική σύνθεση και ιδιότητα. Δεν έχουμε ε, ένα υπόβαθρο που θα ενοποιεί όλα αυτά τα θεσμικά όργανα και θα τα κάνει να δρουν ως μία μονάδα. Για να δούμε τα διάφορα μοντέλα. Αν δω τώρα το κυβερνητικό μοντέλο, το μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δω το Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν, αυτό που ανακαλύπτω και θα τους αρέσει στους Γάλλους συναδέλφους, είναι ένα ημιπροεδρικό μοντέλο. Ιδιαίτερα όταν εκλέγεται ή διορίζεται η Επιτροπή αλλά και όταν ορίζονται οι επίτροποι. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν. Το Συμβούλιο ε, διορίζει έναν υποψήφιο, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να τον εγκρίνει. Μοιάζει αυτό με το σύστημα προηγουμένων μοναρχιών και δεν διαφέρει πολύ από την συνταγματική μοναρχία του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουμε την υψηλή εκτελεστική εξουσία που εξαρτάται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το παράδοξο σύστημα που έχουμε είναι ημιπροεδρικό λοιπόν αν θέλετε. Δεν είναι επικεφαλής ε, αρχηγός κράτους ή κομισιόν, αλλά ο προεδρεύον του Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι κάτι ανάλογο του αρχηγού κράτους. Οπότε είναι μάλλον ένα ημιπροεδρικό μοντέλο. Επίσης, το Συμβούλιο έχει έναν ενεργό τρόπο να επηρεάζει τον πρόεδρο της Επιτροπής. Το ξέρουμε αυτό. Είναι σαφές ότι η απλή παρουσία του πρόεδρου της Επιτροπής σε συνόδους του Συμβουλίου ε, ασκεί επιρροή. Και ακούμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, λαμβάνει μέρος σε συνόδους του Συμβουλίου, καμιά φορά επειδή πρέπει, καμιά φορά επειδή θέλει. Σίγουρα όμως όλα αυτά παίζουν ρόλο και ασκούν επιρροή στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Ε, αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε είναι το πρώτο σύστημα όπου έχουμε ένα τέτοιο προεδρικό σύστημα και η Κύπρος ε, και η Χιλή είχε ένα τέτοιο προεδρικό σύστημα, όχι τα ίδια ακριβώς σε κάθε περίπτωση, αλλά με πολλές ομοιότητες. Εμεί τώρα εδώ τι χρειαζόμαστε. Έχουμε μια εναλλακτική στην προεδρική, στο προεδρικό μοντέλο. Μπορούμε να έχουμε και άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής. Αν έχουμε άμεση εκλογή για τον Πρόεδρο, για το αξίωμα του Πρόεδρου της Επιτροπής, αυτό το μοντέλο που δημιουργούμε θα σημαίνει ότι θα είχαμε έναν υποψήφιο για τη θέση ε, του Προέδρου υποψήφιο των κομμάτων. Αν γίνεται άμεσα η εκλογή, θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το σύστημα από το να προβληθούν υποψήφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αν ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται άμεσα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να ε, ανατρέψει τον πρόεδρο αυτόν ή να το, το απαγγείλει κατηγορία. Ε, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά στο Ισραήλ ο πρόεδρος εξελέγει άμεσα με δυνατότητα να τον παραπέμψει με απλή πλειοψηφία το Κοινοβούλιο και δεν λειτουργήσε καθόλου, απέτυχε τελείως. Μην το κάνουμε λοιπόν. Αν θέλουμε άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής πρέπει να δεχτούμε ότι θα πάμε πιο κοντά στο αμερικανικό μοντέλο ως αποτέλεσμα. Και ποιο θα είναι το πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος. Το πλεονέκτημα θα είναι ότι το Συμβούλιο θα προσαρμοστεί στη, στον πραγματικό του ρόλο που θα είναι ας πούμε, το άνω σώμα, η άνω βουλή σε ένα τέτοιο σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα μπορεί να ανταγωνίζεται με έναν Ευρωπαίο Πρωθυπουργό ή Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής που θα είναι άμεσα εκλεγμένος και εδώ πρέπει να προσέχουμε πολύ γιατί αυτή είναι μια άλλη δυνατότητα συνδυασμού. Δεν, δεν θα έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό σύστημα, το οποίο συνεπάγεται πολλά προβλήματα πώς θα έχω με πρωθυπουργό εκλεγμένο μέσα από το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι και ο πρόεδρος της Γαλλίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλλον φολκλωρική είναι αυτή η προσέγγιση και ουτοπική. Θα επρόκειτο για καρικατούρα. Το λέω για να πω ότι δεν θα είναι βιώσιμο, πρακτικό, εφαρμοσιμό αυτό το σύστημα. Ξαναγυρίζω στη βασική δομή αν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται άμεσα. Αυτό βέβαια θα έχει δύο συνέπειες, δύο πολύ ενδιαφέρουσες επιπτώσεις. Η πρώτη θα είναι ότι με το σύστημα αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να έχει λειτουργεί με σύστημα ε, ψήφου μη εμπιστοσύνης για να ανατρέψει την Κομισιόν. Και η δεύτερη επίπτωση είναι ότι το Συμβούλιο θα ε, ε, πάρει τη θέση της Άνω Βουλής και σταδιακά ο πολιτικός του ρόλος διαχρονικά θα μειωθεί. Θα είναι κάτι σαν νομοθετικό σώμα. αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το νομοθετικό έργο το καθ' αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η γερουσία στη ΣΥΠΑ έχει περισσότερες νομοθετικές εξουσίες από το Κογκρέσο. Ε, υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου η Άνω Βουλή έχει περισσότερες νομοθετικές εξουσίες από την Κάτω Βουλή. Αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Αυτό το, το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος το τις βλέπουμε όταν διορίζονται ομοσπονδιακοί δικαστές ή ο πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες καμιά φορά ε, έχει νόημα η ο προεδρος στις ηνωμενες πολιτειες καμια φορα εχει νοημα η γερουσια να έχει περισσότερες εξουσίες από το Κογκρέσο ή την Κάτω Βουλή. Δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Δεν σημαίνει αυτό οπωσδήποτε ότι το Συμβούλιο θα απογυμνωθεί από κάθε εξουσία. Αυτό που θα γίνει είναι ότι διαχρονικά, συν το χρόνο, θα προσωμιάσει περισσότερο το Συμβούλιο προς μια ανοβουλή και αυτή θα ήταν η πιο συνεπής ε, προσέγγιση αν πάμε για το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Προσωπικά η ιδέα των μεμονωμένων ψήφων μη εμπιστοσύνη δεν θα ενοχλούσαν τόσο πολύ σε αυτό το μοντέλο. Γιατί αν έχουμε άκαμπτο διαχωρισμό μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών, και μάλιστα εγώ θα, δεν θα το ήθελα αυτό, αλλά αν συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα ήταν τόσο κακό να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει στο έργο της Κομισιόν με ψήφους μη εμπιστοσύνης για μεμονωμένους επιτρόπους. Αλλά πρέπει να πω ότι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να διασφαλίσουμε εδώ είναι και θα πρέπει να δούμε αν, ποιος θα το διασφαλίσει αυτό το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Πάντως, ο ορισμός των επιτρόπων θα πρέπει να υπόκειται σε μια διαδικασία ακροάσεων ε, και ελέγχου. Υπάρχει, υπάρχει αυτό το σύστημα, έγινε το 2004 και ο Ιταλός Επίτροπος υποψήφιος απερίφθη το 2009 ε, μια βουλγάρα επίτροπος ε, απορρίφθηκε και ήταν αυτή η διαδικασία των ακροάσεων που κατέληξε ότι έπρεπε να φύγουν δύο. Αν ακολουθήσουμε το προεδρικό μοντέλο δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κακό να υπάρχει ψήφος μη εμπιστοσύνης ιδιαίτερα για αυτούς που θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα ψήφου μη εμπιστοσύνη. Εδώ δεν θα ήταν τόσο κακό να υπάρχει. Βέβαια, η μετατόπιση προς το Προεδρικό ε, αποδυναμώνει το Συμβούλιο και ως ένα βαθμό και το Κοινοβούλιο. Αλλά για να το πω ειλικρινά, πιστεύω ότι έτσι όσο έχουν τα πράγματα, αυτή είναι η όλη εικόνα. Να προσέξουμε το εξής κάτι που ανέφερα έτσι ακροθυγώς, αλλά θέλω να μπω σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Η συνταγματική σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι ενδιαφέρον. Είπα συνταγματική σχέση. Αν τη δείτε εξωτερικά, την τυπολογία αυτής της σχέσης, βλέπετε ότι τα συστήματα διακυβέρνησης που υπάρχουν στο συνταγματικό δίκαιο και στην πολιτική θεωρία εν γέννη. Αν δείτε λοιπόν τι αναφέρεται εκεί και τη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια είναι, νομίζω ότι θα μας οδηγούσε στο να δώσουμε μεγαλύτερη επιλογή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέγει επιτρόπους και αυτό μπορεί να επιτευχθεί σχετικά εύκολα εάν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορεί να επιλέγει από μια ομάδα τριών. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που με ανησυχεί τα ομάλα και κάτι που αναφέρεται σε όλα τα κείμενα τα σχετικά. Από το 1979 την μη προναφερθεί σε ημερομηνία. Δηλαδή, το υπερβολικό μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι εννοώ, είναι δυσκολότατο να έχει κανείς ευέλικτη διακυβέρνηση που να μπορεί να διοικεί σωστά αν έχει 28 επιτρόπους. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό, είναι ότι οι Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν χαρτοφυλάκια και τομείς αρμοδιοτήτων ε, γιγαντίου μεγέθους. Ενώ άλλοι επίτροποι, στην ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν χαρτοφυλάκια τα οποία είναι σχεδόν κενά, κενά περιεχομένου. Αυτό καθε αυτό δημιουργεί ε, κάποια ανησυχία στα κάτι μέλη. Τα φέρνει σε δύσκολη θέση. Ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα, το ελλανδικό πρόβλημα αν θέλετε με το δημοψήφισμα. Αν έχουμε αυτό το πρόβλημα με τους 28 επιτρόπους, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να προσπαθήσουμε άπαξ διαπαντός να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ κρατών μελών. Ίσως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μια δυσνόητη αλλά τολμηρή ιδέα. Μια ισορροπημένη λύση όσον αφορά το πρόβλημα που αφορά την αποδοτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λύση είναι εξή κατά την άποψή μου. Κοιτάμε τις συνθήκες τη Αβώνα. Εξετάζουμε την έγκριση των δύο τρίτων και λέμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν επιτρόπους. Όμως σε αδίποτε περίοδο θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο τρίτα των επιτρόπων δεν έχουν χαρτοφυλάκιο. Ένα τρίτο έχει χαρτοφυλάκιο. Δύο τρίτα δεν έχουν. Άρα, αυτό συμμορφώνεται απόλυτα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δύο τρίτα λοιπόν, μάλλον ανάποδα, δύο τρίτα των επιτρόπων έχουν χαρτοφυλάκιο για μία περίοδο της θητείας και ένα τρίτο δεν έχει χαρτοφυλάκιο και θα γίνεται εναλλακτική κυκλική εναλλαγή ε, εκπεριστροφής κατά τη διάρκεια θητεία. Οπότε θα έχουμε ισορροπία μεταξύ μεγάλων μικρών χωρών, φτωχών και πλουσίων, δυτικών, ανατολικών, βορείων, νοτίων και θα είναι καλό το μείγμα. Δύσκολο να ετοιμάσει κανεί έναν κατάλογο. Έχουμε κάνει όμω πολύ πιο περίπλοκα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν είναι ανέφικτο. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όμως είναι το εξή. Έχουμε δύο τρίτα των επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο, δύο τρίτα των επιτρόπων θα είναι ενεργοί επίτροποι και έτσι βελτιώνει την αποδοτικότητα 18 επιτρόπους. Βέβαια δεν είναι και πολύ ελαφριά δομή, αλλά πολύ ελαφρότερη από την παρούσα. Οι άλλοι επίτροποι θα έχουν έδρα στη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως επειδή είναι άνευ χαρτοφυλακίου, θα έχουν το χρόνο αυτοί οι επίτροποι να εξετάσουν ενδελεχέστερα τα διάφορα ζητήματα, έχουν χρόνο να βοηθούν τους συναδέλφους και έτσι τα συμφέροντα των κρατών μελών τους θα λαμβάνονται υπόψη. Κυρίως τον παρόδο. Αυτός δεν είναι άμεσος ρόλος τους, αλλά άξιζε τον κόπο να τον αναφέρουμε. Τα κράτη-μέλη εκείνα των οποίων οι επίτροποι δεν έχουν χαρτοφυλάκιο και αυτά θα μπορούν να εισακούγονται όταν λαμβάνονται αποφάσεις που θα τις επηρεάσουν τις χώρες. Αυτό αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε. Διότι οι συνθήκες λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι αμερόληπτη, ανεξάρτητη και ισχυρή. Διότι αν είναι ανεξάρτητη, ουδέτερη, αμερόληπτη, αλλά δύναμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανένα ρόλο που μπορεί να παίξει. Θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία δηλαδή ότι θα έχουν αποδυναμωθεί εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλοί όμως δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει ισχυρότερο ρόλο, διότι δεν είναι αρκετά ισχυρή και πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι αμερόληπτη και ουδέτερη. Έχουμε δύο δρόμους. Προεδρική κοινοβουλευτική διαδρομή πρώτα απ' όλα, αλλά ας δούμε πρώτα την εσωτερική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τι βλέπουμε. Αμεροληψία και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι αμελούνται τα συμφέροντα των κρατών μελών. Αντιθέτω, λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, τα θεμητά. Εκείνοι που έχουν γράψει για την αμεροληψία και την ουδετερότητα των εκτελεστικών φορέων γνωρίζουν ότι λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συμφέροντα τότε μπορούν οι φορείς να γίνουν αμερόληπτοι. Έτσι επιτυχάνεται μια ισορροπία και μπορεί να λάβει κανείς υπόψη τις διάφορες ανησυχίες σωστά. Εάν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου οι παρόντες επίτροποι, ε, υπάρχουν παρόντες επίτροποι άνευ χαρτοφυλακίου, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια επιρροή, μπορούν να το εξετάσουν οι επίτροποι και έτσι επιλύονται τα ενδεχόμενα προβλήματα. Και οι άνευ χαρτοφυλακίου επίτροποι θα μπορούν να εκτελούν πολλά καθήκοντα που είναι απλώς αντιπροσώπευσης. Καθήκοντα που εκτελούν σήμερα οι Επίτροποι. Επίτροποι που έχουν δύσκολα χαρτοφυλάκια, αλλά πρέπει να εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλοί αντιπρόεδροι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πηγαίνουν σε διάφορε χώρε. Έχουν πάρα πολλού ρόλου που πρέπει να παίξουν, που δεν σχετίζουν απαραίτητα με το χαρτοφυλάκιό του, αλλά πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά του που είναι η θεσμική εκπροσώπηση. Και αυτού του είδου η εκπροσώπηση, τα ταξίδια στα διάφορα κράτη με τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι κάτι που θα τα κάνουν οι άνευ χαρτοφυλακοί επίτροποι. Και θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του του τον τρόπο. Αυτή είναι μια πρόταση. Μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Διάκριση μεταξύ επιτρόπων μετά χαρτοφυλακίου και εκείνων άνευ χαρτοφυλακίου. Και κλείνοντας, διότι ήδη μακρηγόρησα κάπω με την παρουσίαση μου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι έχουμε και δύο-τρία τεχνικής φύσου ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα θέματα ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα εν γέννη. Είναι πιο σεξι θα έλεγα σαν ζητήματα. Και αφορούν μακροσκοπική θεώρηση των πραγμάτων. Αλλά είναι αρκετά αυτά ε, κρύβονται αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες και αφορούν την ισορροπία δυνάμων μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου βέβαια, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό σε αυτή τη φάση. Αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες λοιπόν καμιά φορά ε, είναι το ζουμί. Ενώ ε, έχουμε και τους δούριους ύπους διαφόρων μακροσκοπικών πτυχών. Λοιπόν, κάτι που θεωρώ ότι ήδη ανέφερα, αλλά πρέπει να επανεξεταστεί, είναι και το εξής. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εσωτερικεύσει την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ειλικρινά ότι τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα εδώ. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει ή να απορρίπτει συμφωνίες είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Είχαμε και το προηγούμενο τη συμφωνία SWIFT. Είτε κανεί συμφωνεί με τη θέση που ελήφθη την πρώτη φορά που απερίφθη η συμφωνία SWIFT, παρόλα αυτά αυτό απέδειξε πολύ καλά ότι έχει δύναμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι μπορεί να απορρίψει συμφωνίε που έχουν υπογραφεί, διεθνεί συμφωνίε. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε και μια άλλη ιδέα. Δηλαδή, ότι τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θεωρούν ότι πρέπει να συνοδεύουν όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ότι οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν στις των διεθνών αυτών διαπραγματεύσεων. Ειλικρινά αυτό πιστεύω ότι είναι λανθασμένο. Άλλο η συνοδεία, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον τελικό λόγο κατά πόσο τα κείμενα που εγκρίνονται κατόπιν διαπραγματεύσεων εγκρίνονται είτε απορρίπτονται. Άρα είναι σημαντικό να παρακολουθούνται και να συνοδεύονται οι διαπραγματεύσει. Όμω δεν νομίζω ότι αυτό που αποκαλούσε ο Τζον Λοκ ομοσπονδιακή εξουσία στο κείμενό του θα πρέπει να ε, υπησέλθει εδώ. Δηλαδή ότι η μη εκτελεστική εξουσία έχει το δικαίωμα τη διαπραγματεύση όσον αφορά τη Διεθνή Συμφωνία. Δικαίωμα έγκρισης ή κύρωσης είναι κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωση του Σέγγεν και εκεί έπρεπε να δεχτούμε ή να απορρίψουμε συμφωνίες και έγιναν απόπειρες περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού του Κοινοβουλίου από τη διαδικασία. Νομίζω ότι η συμφωνία SWIFT και άλλες παρόμοιες έδειξαν πώς μπορεί να συνοδεύει το Κοινοβούλιο και να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις εκ του μακρόθεν. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποτελεσματικά συμμετάσχει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κοινοβούλιο, εθνικό κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κατάφερε, έχει καταφέρει να έχει λόγο, ακόμα και αν δεν το κάνει πάντα επισήμως. Τι είναι να κινείται περισσότερο από ότι τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό ε, δεν είναι κάτι που αμφισβητείται και θα, ούτε πρέπει να αμφισβητηθεί, διότι καμιά φορά τα εθνικά κοινοβούλια δεν ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει εκτός συνόρων, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπερεθνικό χαρακτήρα εξορισμού. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι πολύ πιο καλά εστιασμένο στις διεθνείς συμφωνίες. Άρα είναι κατανοητό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμμετέχει. Νομίζω, λοιπόν, ότι με τις διεθνείς επιτροπές που έχουμε στο Κοινοβούλιο πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει το ρόλο του ε, θετικού διαμεσολαβητή στις συζητήσεις, κυρίως αν συμμετέχουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και το άλλο θέμα, δηλαδή πώς διευθετούμε ζητήματα που άπτονται της Διοργανικής Συμφωνίας. Διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία πλαίσιο στις αρχές αυτής της θητείας Πρέπει να γνωρίζουμε τώρα κατά πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την διοργανική συμφωνία. Μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσει, Πρέπει να γίνουν ακροασει για τους επιτρόπους κλπ. κλπ. Συμφωνούμε όμω όσον αφορά τις βασικές γραμμές δράσης. Πιο κοινοβουλευτική προσέγγιση, πιο προεδρική προσέγγιση. Θέλουμε ενισχυμένο ρόλο της, ε, του προεδρικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όχι. Καμιά φορά όταν υιοθετούμε το προεδρικό μοντέλο αυτό ίσως θα οδηγούσε συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε και ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε ξεκάθαρη άποψη δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο πραγματικά θα συμφωνήσει με τη δική μας άποψη που εκφράζεται συμφωνία πλαίσιο. Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο επίτευγμα για μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως πιστεύω ότι τίνει περισσότερο προς το να αφήνει αυτές τις συμφωνίες να εκπνέουν και πάντα προέβαλε αντιστάσεις στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις συμφωνίες πλαίσιο. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ε, προσέχουν όλος ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό αλλά επεδείχθη μεγάλη ευελιξία και βιασύνη καμιά φορά καμιά φορά υπερβολική βιασύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ταχεία σύναψη συμφωνιών στην πρώτη ανάγνωση άτυποι τριμερείς διάλογοι έχουν πραγματοποιηθεί κλπ. Πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απεμπολίσει τα αιτήματά του στην ε, προσέγγιση αυτή για να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσει να ξεπεράσει τους επίσημους κανόνες να υπερκεράσει τους επίσημους κανόνες του τριμερούς διαλόγου. Καταλαβαίνω ότι το ανεπίσημο μοντέλο είναι ελκυστικό, όμως ανησυχώ για το που πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Καμιά φορά λοιπόν, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η νομοθεσία, ίσως προχωράμε προς κατευθύνσεις που ευνούν περισσότερο τις ανεπίσημες διαδικασίες, ίσως σε υπερβολικό βαθμό. Όλα κινούνται αργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι περίπλοκα κατά όργανα που συμμετέχουν στις διαδικασίες. Όμως, αν δούμε τη γερμανική νομοθετική διαδικασία, το γερμανικό σύστημα, βλέπουμε ότι εκεί υπήρχε μια μεγάλη τάση το 94, το 95 και τα επόμενα έτη να υπάρχουν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις, να πραγματοποιούνται διαργασίες ανεπισήμως. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνταγματική ανεπίσημη νομοθετική διαδικασία. Προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από άκαμπτες δομές. Όμως πιστεύω ότι καμιά φορά αυτό σημαίνει ότι εξαρτούμεθα του δικαιωματο ελέγχου που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ίσως οι συνάδελφοι να μην ικανοποιούν αυτή την ιδέα. Όμως ίσως θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε το ρόλο της Ολομελίας του Κοινοβουλίου με τις Επιτροπές του Κοινοβουλίου. Η παραδείγματι, όταν οι συνάδελφοι παρουσιάζουν εκθέσεις τους και η έκθεση μετά απορρίπτεται στην Ολομέλεια, λέγουν αυτοί αυτό είναι κάτι που εγκρίθηκε στην Επιτροπή με 20 ψήφους παραπάνω. Και αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε απογοητεύσεις για τους συναδέλφους. Νομίζω λοιπόν ότι η κυριαρχία και η επικράτηση των επιτροπών έναντι τη Ολομέλειας είναι κάτι που θα μπορούσε να μας οδηγήσει και σε δυσκολίες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαι όσο πιο ευέλικτη γίνεται, όμως θα πρέπει να διατηρηθούν οι επίσημες διαδικασίες, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου. Και κάτι άλλο Πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαμαρτύρεται και σωστά πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι προκύπτουν προβλήματα όταν θέτουμε ερωτήματα. Έχουμε συναδέλφους σε διάφορες αντιπροσωπείες οι οποίοι θέτουν εκατοντάδες ερωτήσεων με το σύστημα copy-paste του υπολογιστή. Βασικά ρωτούν την ίδια ερώτηση από την οπτική γωνία του κάθε κράτους μέλους όμως. Και αυτό ε, απλώς αυξάνει τα στατιστικά στοιχεία για τις εργασίες κάθε εβδομάδα και προσπαθούν να δείξουν ότι έτσι εκπροσωπείται κάθε χώρα σωστά και αυτό είναι δαπανηρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοστίζει περίπου 5.000 ευρώ. Παρόλο λοιπόν που είναι οδυνηρό αυτό που λέω για μένα, ίσως αυτή η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που θα πρέπει να συγκρατηθεί αυτή η σημαντική χρήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οδηγεί σε κολλησιεργία όσον αφορά μια έκθεση και ίσως ε, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε από μια πειθαρχική σκοπιά. Ίσως να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία κυρίων για να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν προς όφελός μας. Και κάτι άλλο το θέμα των νομοθετικών πρωτοβουλειών, το αιώνιο ερώτημα, πάντα το συζητάμε αυτό. Η συμφωνία πλαίσιο μας έκανε να προχωρήσουμε αρκετά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, μας επέτρεψε κάποια επιρροή και δικαίωμα πρωτοβουλίας, δικαίωμα πρωτοβουλίας ακόμα και πριν ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει το δικαίωμα του πρωτοβουλίας ε, αχαλήνοτα και η αποδύναμωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε παρατηρήσει ίσως είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. Νομίζω ότι η ιδέα της ενίσχυσης των νομοθετικών πρωτοβουλίων του Κοινοβουλίου δεν είναι απαραίτητα μια σωστή ιδέα και νομίζω ότι σωστά διατείνεστε ότι ο αδύναμος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει συμπιεστεί μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι κάτι που βοηθά και θα αποδυναμωθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν παραμείνει σε αυτή τη θέση κολλημένη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να ενισχύσουμε το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε ίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ασκήσει το πλήρε δικαίωμα που έχει για νομοθετική πρωτοβουλία. Και ίσω θα, θα έπρεπε να μειώσουμε τη δική μας ε, εξουσία όσον αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία δεόντως. Και μετά, η συνθήκη της Αβώνας ε, που αποδίδει διάφορες αρμοδιότητες. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ εφαρμοστικών πράξεων και εξουσιοδότηση πράξεων και να μην υπάρχει χειραγώγηση σε αυτόν. Από ό,τι που έχουμε δει είναι, για να το πούμε ειλικρινά, συστηματική κατάχρηση αυτών των εργαλείων από πλευράς Συμβουλίου, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να έχει δυσκολότερο ρόλο και να δυσκολεύεται και ο ρόλος ε, που έχει το Κοινοβούλιο για την άσκηση ελέγχου. Αυτές οι καταξισοδότηση πράξεις και εφαρμοστικέ πράξεις δεν μπορούν συνεχώς να συγχωνεύονται όπως γίνεται συχνά κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ουσιαστικά λοιπόν η ιδέα σύμφωνα με την οποία εμείς θα πρέπει να εστιαστούμε επί ανάθεση σε κατεξοδότηση πράξεις αποφάσεων που είναι πολιτικής φύσεως είναι κάτι που το σκεφτούμε. Το γερμανικό και ιταλικό μοντέλο μας δείχνει ότι αυτό που έχει πολιτική ουσία πάει στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε κατεξοδότηση πράξης. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε τι είναι ουσιαστικό και αυτό πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ εφαρμοστικών πράξεων και κατεξοδότηση πράξεων. Όμως, εάν ελέγξουμε τις κατεξοδότης συμπράξεις αποτελεσματικότερα χρησιμοποιώντας το άρθρο 190 για τη συνθήκη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διάφορες άλλες ισχύουσες ρήτρες, παραδείγματο χάρη αν συμπεριλάβουμε δεσμευτικές οδηγίες στο βασικό κανονισμό που θα ορίζει πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί και πότε δεν μπορεί να υιοθετεί κατεξοδότηση πράξης και ούτω, και καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διάφοροι συναφείς φορείς μπορούν να εμπλακούν στην προετοιμασία των κατεξοδότησης πράξης, πράξεων μάλλον. Όλα αυτά είναι τιτάνιο έργο, δεν μπορούμε να αναμειχθούμε σε όλα. Αλλά να σας υπενθυμίσω τις βασικές μου ανησυχίες ήθελα. Και δουλειά μου τώρα θα είναι να συναθροίσω τις συνεισφορές των συναδέλφων Όλα όσα που είναι συνάδελφοι θα είναι χρήσιμα, είμαι βέβαιος γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε παραλήψεις ή κενά της παρουσιάσεώς μου και θα μπορέσετε να μου βοηθήσετε ενδεχομένω να βρω κάποια διέξοδο, κάποια πορεία για το μέλλον όταν ετοιμάσω το αρχικό μου κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ή κάνατε πραγματικό μάθημα συνταγματικού δικαίου ευρωπαϊκού. Σας ευχαριστούμε. Εξετάσατε όλες τις πτυχές όλες το λεπτομέρειες του προβλήματος που απαιτεί ουσιαστική ενδελεχή ανάλυση για να γίνουν επιλογές. Σας ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο σε εκείνον που θα θέλει να μιλήσει. Ο συνάδελφος Ντάφ, συγγνώμη, είναι εκείνος που ζήτησε το λόγο πρώτος. Well, I... Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Παύλο Ραντζέλ αλλά και τους ε, διερμηνείς για τη δουλειά που έκαναν πρέπει να προσέξουμε να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στα πλαίσια της εντολής της Επιτροπής μας. Δηλαδή, την εφαρμογή των συνθήκων σύμφωνα με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αρκετά ευρύ το θέμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τίθενται σημαντικά θεσμικά ερωτήματα και συνταγματικά. Ο εισηγητής ανέφερε πολλά από αυτά, αλλά αν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που να χρησιμοποιηθεί και από το επόμενο κοινοβούλιο, να είναι χρήσιμη για το επόμενο κοινοβούλιο, πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη πειθαρχία, αυτοπιθαρχία. Και αυτό πώς ακριβώς από τη συνθήκη της Λισαβόνας επωφελήθηκε το Κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε τις νέες του δικαιοδοσίες σωστά, με κάποια επιτυχία, Τώρα για το διορισμό της Επιτροπής εμείς δεν ξέρουμε ποιε ακριβώς θα είναι οι συνέπειες της αλλαγής της συνθήκης ως προς τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν πριν να το δούμε στην πράξη. Το θέμα δεν είναι απλώς η δυνατότητα ή η ικανότητα των πολιτικών ομάδων και κομμάτων να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες τους, αλλά και το κατά πόσον ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κομισιόν που θα έχει περισσότερη νομιμοποίηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά πόσο λοιπόν θα μπορέσει να επηρεάσει το διορισμό των υπολείπων επιτρόπων περισσότερο από ό,τι οι προηγούμενοι. Θα με ενδιέφερε πολύ η πρόταση του Παύλου Ράντζελ να ξαναεξετάσουμε την δομή, τη λειτουργία της Κομισιόν και τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να οργανώσει, για να το πω έτσι, καλύτερα την δομή αυτή από ό,τι μέχρι τώρα. Πιστεύω όμως όπως λέει και το σύνταγμα που προέβλεπε η ομάδα Σπινέλη ότι σύντομα πρέπει να παρατήσουμε πλέον την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει ένας επίτροπος τουλάχιστον για κάθε χώρα. Ήταν σωστό νομίζω που προβλέφθηκε ότι πρέπει να μειωθεί το μέγεθος της Κομισιόν και ότι λάθος θα ήταν να επιβληθεί στο Συμβούλιο η ευθύνη να βρει έναν τρόπο, έναν τύπο καλύτερης ή πιο δίκαιας εναλλαγής μεταξύ των χωρών μελών. Αυτό ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Αυτό το έλεγα από την αρχή και αποδείχτηκα σωστός. Πέραν των άλλων είναι φανερό ότι ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνος αποδυναμώθηκε κυρίως η Κομισιόν ιδιαίτερα σε σύγκριση με το Συμβούλιο. Και αυτό δεν είναι καλό για την Ένωση, να είναι αδύνατη η Επιτροπή δηλαδή. Αντίθετα προς το συμφέρον της θα ήταν να αλλάξει, να μεταμορφωθεί η Κομισιόν από αυτό που είναι σήμερα σε πραγματική κοινοβουλευτική κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και στοιχεία και άλλα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι γιατί ο εισηγητής ανέφερε το ρόλο των κοινοβουλευτικών επιτροπών ως προς την Ολομέλεια τις εσωτερικές μεθόδους λειτουργίας πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι λειτουργίες μας και έως προς τους τριμερείς διαλόγους για να διασφαλίσουμε τις βελτιώσεις που μας έδειξε η εμπειρία ως προς τη διαδικασία έγκρισης της Κομισιόν ας πούμε και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια συμφωνία πλαίσιο. Και όπως λέει ο συγητής πρέπει νομίζω να προσπαθήσουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο να είναι και αυτό μέρος της διαθεσμικής συμφωνίας, της συμφωνίας πλαισίου με το Κοινοβούλιο και ως προς την κατάρτιση του προγράμματος της Επιτροπής της Κομισιόν. Είτε του αρέσει είτε όχι πρέπει να συμμετάσχει το Συμβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Αμφισβητώ βέβαια το, το ρόλο του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Είναι και αυτό ένα θέμα. που απαιτεί έκθεση. Πρέπει να ενδυναμωθεί η εντολή που έχει το Κοινοβούλιο για τις ερευνητικές επιτροπές και βεβαίως πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην συμπλήρωση του καθεστώτος για τα πολιτικά κόμματα. Χωρίς αυτό το ουσιώδες δημοκρατικό στοιχείο ε, έχουμε μεγάλες αδυναμίες στο Κοινοβούλιο και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό όταν θα προετοιμάζουμε το έδαφος για την επόμενη θητεία. Αναμένω βέβαια το σχέδιο έκθεσης και είμαι βέβαιος ότι τότε θα έχω και άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Ο κύριος Μορέιρα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την ευρύτατη επισκόπηση των συνταγματικών πτυχών της σχέσεως ε, Κομισιόν Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως, το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο περιορισμένοι όσον αφορά την εντολή, δηλαδή το θέμα που θα καλύψει αυτή η έκθεση. Από ό,τι φαίνεται, το πεδίο κάλυψης της εκθέσεως αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε απόλυτα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ερώτηση λοιπόν. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε με τον εισηγητή ή όχι, θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά τα σημαντικά θέματα της, ε, της συνταγματικής μορφής που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Είναι σωστή στιγμή, η σωστή ευκαιρία αυτή να το κάνουμε αυτό. Εγώ θα προτιμούσα να περιοριστούμε λίγο περισσότερο και να εστιαστούμε επί του πυρήνα του ζητήματος. Θα προτιμούσα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό τι αλλαγέ που επιφέρει η συνθήκη της Μπορεί να το κάναμε αυτό, το πετύχαμε. Ε, μπορούμε να δούμε ποιε είναι θεσμικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ άλλαξαν αυτέ οι σχέσει μετά τη συνθήκη της από πλευρά νομοθεσία, διεθνών συμφωνιών και πολιτικών διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινούσα εγώ όσον αφορά την ε, επισκόπηση της προόδου που επέφερε η συνθήκη της Σαβόνας και να δω ποιοι τομεί θα μπορούσαν να βελτιωθούν όσον αφορά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της ε, Διεθνής Συμφωνίας. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά πόσο κάναμε αυτά που αναμενόταν μετά τη συνθήκη της Σαβόνας και ίσως να υπογραμμίσουμε κάποια κενά, κάποια προβλήματα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε τελικά αλλά και όσον αφορά τις ε, βελτιώσεις όσον αφορά τα προβλήματα που εντοπίσαμε και να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση στο μέλλον, τούτων λεχθέντων. Εγώ θα επέλεγα τρεις τομείς. Πρώτον, νομοθετικό τομέας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι καταφέραμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, τη δυνατότητα να ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν, για το ποιους νομοθετικούς τομείς θα θέλαμε να εξεταστούν. Αυτό είναι πραγματικά μία πρόοδος. Πιστεύω επίσης ότι η κανονική νομοθετική διαδικασία είναι τεράστια βελτίωση εν συγκρίση με τις όλες τις διαδικασίες. Έχω κάποιες αμφιβολίες, περισσότερες αμφιβολίες όσον αφορά τις κατεξοσοδότηση πράξης και τις εφαρμοστικές πράξεις. Μέχρι τώρα ε, το να ευθυγραμμίζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο με τις επιταγές ηθίξης της Αβώνας όσον αφορά τις εφαρμοστικές και τις κατεξιδότητες συμπράξεις είναι κάτι που παραμένει ατελές. Τόσα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο φέρει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς. Και είναι λυπηρό το ότι δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε όσον αφορά τις κατεξουσοδότησης πράξεις. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με την ε, θέση σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αυτή είναι η ισχύουσα άποψη, η επικρατούσα άποψη. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Αν υπερφορτώσουμε τις ε, νομοθετικές διαδικασίες μέσω ειδικών ψηφοφοριών για τεχνικά ζητήματα και επιβαρύνουμε όλος ιδιαίτερο τα διάφορα νομοθετικά βήματα, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πάρα πολύ συχνά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να δίνουμε κατά εξουσιοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο πρόσφατο παράδειγμα μπορούσα να παραθέσω ήταν η οδηγία για τις ιατρικές συσκευές που εμπεριείχε κανονισμούς με τόσες τεχνικές λεπτομέρειες 98% των μελών δεν καταλάβαιναν ακριβώς περί τίνος επρόκειτο και τι εψήφιζαν. Θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό εκ των προτέρων να είχαμε θεσπίσει κάποιους γενικούς κανόνες βάσει πολιτικών ε, κριτηρίων όπως ανέφερε ο κ. Ρανζέλ και με βάση αυτά τα κριτήρια θα ανελάμβανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά που είπα για το συγκεκριμένο κανονισμό ισχύουν και για πολλούς άλλους. Εάν εγκαταλείπαμε τις προκαταλήψεις μας και την καχυποψία μας έναντι των κατεξοδότησης πράξης ε, ε, ε, θα μπορούσαμε να περισσότερο επί των βασικών πολιτικών μας προτεραιοτήτων και νομοθετικών προτεραιοτήτων. Ήδη ελέγχουμε τις κατεξοδότηση πράξεις. Αυτό αναφέρεται σαφώς στη συνθήκη και συμπεριλαμβάνεται και στη διοργανική συμφωνία. Και όσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις, νομίζω ότι ίσως να αφησυχάσαμε υπερβολικά οι κανόνες περί επιτροπολογίας έχουν κενά. επιτρέπουν γενικόλογες εφαρμοστικές πράξεις που φαίνεται να είναι σχήμα οξύμορων. Αν είναι μια εφαρμοστική πράξη θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεκριμένη και ειδική. Όταν είναι κάτι γενικό θα πρέπει να αφορά νομοθετική πράξη ή κατεξουδότηση πράξη. Πιστεύω ότι η κατεξουσιοδοτηση πραξη πιστευω οτι η εξαιρεση που έχει μπει στην επιτροπολογία μέσω των εφαρμοστικών πράξεων αποτελεί δικείμενο κατάχρησης. Έχουμε φυσικάσει υπερβολικά σε αυτό το τομέα. Έχουμε επιτρέψει εφαρμοστικέ πράξεις να χρησιμοποιούνται που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μόνο τα κράτη-μέλη ελέγχουν τι εφαρμοστικές πράξεις. Πολλά μπορούν να γίνουν εκεί, σε αυτό το μέτωπο. Ούτω ώστε να υπάρξει σαφής διαχωριστική γραμμή όσον αφορά την χρήση των εφαρμοστικών πράξεων και των κατασκευοδότησης πράξεων και θα πρέπει να είμαστε λιγότερο διστακτικοί όσον αφορά την χρήση των κατεξοσοδότησιν πράξης και ακόμα πιο διστακτικοί όσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις. Σχετικά με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, πολύ συχνά ονομαστικές ψηφοφορίες επί δωδεκάδων τροπολογιών ε, που είναι πάρα πολύ τεχνικές και πάρα πολύ λεπτομερείς, αυτό είναι κάτι που θα γινόταν καλύτερα στις επιτροπές. Πολύ συχνά περνάμε μισή ώρα ψηφίζοντας δεκάδες επί δεκάδων νομοθετικές τεχνικές λεπτομέρειες και αυτό δεν είναι, αποτελεί την καλύτερη χρήση του χρόνου μας. Αν τα μέλη, αν το κοινό παρακολουθούσε τις ολομέλειες δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Θα λέγανε ότι περνάνε το χρόνο τους με τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν θα ενδιέφερε το κοινό καθόλου και τα ίδια τα μέλη δεν έχουν σαφή άποψη επί πολλών σημείων που ψηφίζουν. Θα ήταν πιστεύω πολύ πιο καλό, καλύτερη προσέγγιση όλα αυτά να εξετάζονται ε, εις βάθος στις διάφορες αρμόδιες επιτροπές. Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία η συνθήκη της ε, Λισαβόνας έδωσε νέες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσει με διεθνείς συμφωνίες, για να εγκριθούν οι διεθνείς συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποια επιρροή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κάτι που δεν θα είχε διαφορετικά. Υπάρχουν δύο πολύ κρίσιμα σημεία στον τομέα αυτό. Πρώτα απ' όλα, κάτι που ανέφερε και ο συγκητής, η συμφωνία SWIFT, που απερίφθη από το Κοινοβούλιο στην αρχή. Η δεύτερη συμφωνία SWIFT απετέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεως στην συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το Κοινοβούλιο πήγε στη Ουάσιγκτον και διαπραγματεύτηκε, συμμετείχε στη διαπραγματεύση για βασικά σημεία ε, ε, τη SWIFT 2. Ήταν και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο εκεί. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών και θα πρέπει να έχουμε να, αυτά τα παραδείγματα όπως το SWIFT να μην είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. Όσον αφορά την Κολομβία και το Περού που νομίζω ότι αναφέρθηκαν σαν χώρες τις οποίες τα κοινοβούλια συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις πριν από την κύρωση συμφωνιών η Κολομβία και το Περού και στην Κολομβία και στο Περού συμμετέχουν τα κοινοβούλια στις διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν εγκριθούν. Τα κοινοβούλια ε, καθορίζουν έναν οδικό χάρτη, την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και το κοινοβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία στην ολομέλειά του. Αλλά και αυτό ε, ήταν Είχαμε και εκεί εξαιρετική ε, περίπτωση όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι διαπραγματεύσει με αυτέ τι χώρε. Όσον αφορά το να συνοδεύει το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό τη Εθνή Συμφωνία, η εμπειρία μα ήταν καρποφόρα και επικοδομητική κατά το παρελθόν. Δουλειά μα είναι να παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν, να συλλέγουμε πληροφορίε ε, για τι συζητήσει και τι διαπραγματεύσει και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ πιο θετική, σε πιο πλεονεκτική θέση από τα Εθνικά Κοινοβούλια το κάνουμε αυτό. Πολύ συχνά απλώ τυπικά επικυρώνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια τι συμφωνίε. Εμεί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Η εμπειρία μα δείχνει ότι αυτό είναι κάτι αξιέπαινο. Και χάρη σε εμά, πιστεύω, πολλά στοιχεία συμπεριελήφθησαν στι συμφωνίε κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Παραδείγματο χάρη, στο δικό μου τον τομέα υπάρχουν πολλέ διεθνεί συμφωνίε για το διεθνέ εμπόριο και αυτό που έχουμε ε, δημιουργήσει εδώ είναι καλή πρακτική. Και το παράδειγμα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου είναι κάτι που να ακολουθήσουν και άλλες επιτροπές. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι στις διεθνείς εμπορίες. Δηλαδή, ο χρόνος μεταξύ συνάψου συμφωνίας και θέση σε ισχύ μια συμφωνίας. Μπορεί να περάσουμε και τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια καμιά φορά, πέντε χρόνια. Γιατί, διότι στο τέλος των διαπραγματεύσεων, όταν η συμφωνία υποβληθεί στο Κοινοβούλιο, χρειάζεται μέχρι ένας χρόνος για να μεταφραστεί αυτή η συμφωνία. Και, για, και να ελεγχθεί από πλευράς νομικής. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Είναι λυπηρό αυτό, διότι υπάρχουν συμφωνίες που είναι πολύ επωφελείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στον τομέα του εμπορίου, αλλά χρειαζόμαστε δύο, τρία και τέσσερα χρόνια μέχρι ότου να τεθούν σε ισχύ συμφωνίε αυτέ. Σε κάποιε περιπτώσει πρέπει προσωρινά να τεθούν σε ισχύ. Άρα πρέπει να είμαστε φάνταστοι και δημιουργικοί όταν περιμένουμε για την έγκριση ή κύρωση των διεθνών συμφωνιών από κοινοβούλια. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στον πολιτικό έλεγχο επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, μπορούν και θα έπρεπε να βελτιωθούν. Ήδη έχουν βελτιωθεί. Και αρκετοί συνάδελφοι έχουν δει ότι μπορούν να βελτιωθούν και οι λειτουργίες των διαφόρων επιτροπών το Κοινοβούλιο έχει κερδίσει νέες εξουσίες ελέγχου επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε σημειώσει πρόοδο να αλλά πολλά πρέπει και μπορούν να γίνουν ακόμα. Όμως, εν τέλει, πρέπει να αναφέρω ένα στοιχείο στο οποίο υπολοιπόμεθα των προσδοκιών. Και αυτό είναι κάτι που ανέφερε ο κ. Νταφ, δηλαδή την ομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα. Οποιοςδήποτε που ακολουθεί κοινοβουλευτική προσέγγιση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμού συμπεριλαμβανομένου, δεν θεωρώ ότι είμαι υπέρ της προεδρική προσέγγισης και ο κύριος ε, Ρανοζέλ το ξέρει αυτό, συνάδελφός μου. Ξέρουμε ότι καμία κίνηση προς κοινοβουλευτική προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί εκτός εάν παγιωθεί και εδρεωθεί ο ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αυτό έπρεπε να είχαμε κάνει από την αρχή της θητείας μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Ισαβώνας. Προσπαθούμε, προσπαθήσαμε να διαβρύνουμε το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και αποτύχαμε σε ένα βασικό σημείο εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αυτό δεν μπορεί να λείπει από τη σχετική έκθεση που αφορά το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, κύριε Μορέιρα, για μια παρέμβαση που συνέβαλε ε, με σημαντικό τρόπο στη συζήτηση αυτή. Ο κύριο Σόλτ έχει ζητήσει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Νταφ. γιατί παρακολούθησα με πολύ ενθουσιασμό, προσδοκίες, ε, την έκθεση, όπως και ο συνάδελφος Νταφ και όταν ε, κατατεθεί θα πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος για να αναλύσουμε πολλές όψεις που ανέφερε ήδη ο εισηγητής. Ευχαριστώ για την ε, ανταλλαγή απόψεων που επέτρεψε αυτό. Πρέπει όμως να το δούμε πιο πολιτικά το θέμα. Εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω δύο θέματα που πιστεύω ότι θα έχουν κεντρική σημασία. Ε, προκειμένου να αναφερθεί, να στηριχθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας η έκθεση και να δείξει τις δυνατότητες για το μέλλον. Ε, εμείς ε, συζητούμε την έκθεση σε συγκεκριμένη πολύ σημαντική ιστορική στιγμή. Η κόποση από την Ευρώπη, ο ευρωσκεπτικισμός αυξάνονται και στα κράτη-μέλη όλα γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Και οι επόμενες εκλογές στο Μάιο θα δείξουν ότι αν δεν μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή τη βασική προβληματική, πώς μπορούμε δηλαδή να ε, έχουμε θεσμικά όργανα που να λειτουργούν βάσει της συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη με ρεαλισμό τα προβλήματα των ανθρώπων και να τα λύνουν με τρόπο πολιτικό, τότε θα αποτύχουμε στο εγχείρημά μας. Και νομίζω αυτή είναι η βασική πολιτική διάσταση της έκθεσης που πρέπει να αναδείξουμε. Δεν θέλω δηλαδή να μιλάμε για τους τύπους και για μηχανισμούς και σχέσεις ε, ε, μηχανικές και μηχανιστικές μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Μιλάμε αντικειμενικά για τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι ε, σωστές. Το Συμβούλιο δεν θέλει να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί, γιατί η θέση ισχύω. των άλλων θεσμικών οργάνων ε, και η ανάγκη για αύξηση εξουσιών καταδεικνύουν μια υπερβολή στο κομμάτι του Συμβουλίου. Και νομίζω ότι εκεί Πρέπει να δείξουμε περισσότερο θάρρος και εμείς και ο εισηγητής για να αναδείξει αυτές τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλιώς ε, θα είναι μια έκθεση επιφανειακή η οποία ε, αναφέρεται σε τρόπους λειτουργίας μηχανιστικά και υποβάλει σχετικέ προτάσεις. Την ουσία του προβλήματος όμως δεν θα την έχουμε πιάσει, γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο θάρρος στην έκθεση αυτή. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι το εξή. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ε, σε πολλά θέματα που αναφέρονται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Πώς οργανώνεται ε, μέσα από την ε, δραστηριότητα ελέγχου πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Χρειάζεται όμως και το νομοθετικό δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να καταδεικνύουμε τα σημεία που χωλένουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε, παίρνουμε πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα, να έχουμε σε βασικά θέματα δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας, ότι εδώ πρέπει να βελτιωθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, και ε, πολύ σημαντικό είναι το πολιτικό βάρος που ε, έχει κάθε θεσμικό όργανο και στη σχέση μεταξύ τους. Τέλος, θα πρέπει να διατηρηθεί ο ρόλος των βουλευτών και να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των πολιτικών ομάδων. Δεν πρέπει να περιοριστούμε δηλαδή στο να εξετάσουμε μόνο το έργο των επιτροπών. Πρέπει να είναι πολιτικό το κοινοβούλιο και να μπορεί να ανοίγει νέους δρόμους προς την ολοκλήρωση. Και γι' αυτό χρειάζονται οι πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές. Χρειάζονται βεβαίως οι ακροάσεις, οι γραμματείες, οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Ε, όλα αυτά χρειάζονται. Είναι το νομοθετικό έργο του ε, Κοινοβουλίου. Το διασφαλίζουν. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε πού χρειάζονται κατεξουσιοδότηση πράξης, πού θα εφαρμοστούν εκτελεστικές πράξεις, πώς θα ορίζονται οι... πώς θα ορίζεται το έργο των επιτροπών κλπ αλλά βασικό είναι να δούμε ε, τις πολιτικές δομές που υπάρχουν. Τέλος, για θα σταματήσω με αυτό, πρέπει να δούμε ε, τη θέση του Κοινοβουλίου και της πολιτικής που γίνεται εδώ και πώς όλα αυτά θα συνδεθούν με, πιο ε, στέρεο τρόπο με την κοινωνία. Πολλές φορές ε, πράγματι το είπαμε ότι ε, είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα. Και εμείς φταίμε γι' αυτό γιατί δεν κάνουμε διάφανη την πολιτική. Δεν λέμε δηλαδή σε ποιο επίπεδο ε, αναφερόμαστε ή ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος είναι υπόλογος για κάθε θέμα. Αν τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, πού είναι αρμόδιο το Συμβούλιο, πού τα κράτη-μέλη, πού ισχύει η επικουρικότητα, πού πρέπει να παρεμβαίνουμε, τότε θα βελτιωθούν πολύ τα πράγματα και δεν θα χρειάζεται να φοβόμαστε ότι κάνουμε μια πολύ συγκεντρωτική Ευρώπη. Γιατί θα μπορούμε να πούμε ότι κάποιες ε, εξουσίες θα δοθούν σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. Και όχι μόνο το ευρωπαϊκό. Υπάρχει αυτή η διαδική σχέση μεταξύ λήψης αποφάσεων σε επίπεδο κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο καλό θα ήταν να προσπαθήσει η έκθεση να το καταγράψει και να αναφερθεί εδώ στην εμπειρία του SWIFT και άλλων συμφωνιών. Γιατί έτσι θα ξεκαθαριστεί πού στις διεθνείς συμφωνίες ε, θα πρέπει να ε, απλουστεύσουμε τις δομές λήψης των αποφάσεων για να μην περνάει τόσος χρόνος ε, από την σύναψη μιας ε, διαδικασίας και τη θέση σε ισχύ του. Να, μειώνουμε, να μειώσουμε ε, το διάστημα που περνάει, γιατί πολλές φορές σε μια θητεία συζητείται ένα θέμα και στην επόμενη θητεία αρχίζει να τίθεται σε εφαρμογή και να αλλάζει και να επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Αυτό πρέπει να γίνεται πιο σύντομα. Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και ευθύνες της δικής μας της Επιτροπής. Να δράσουμε ενισχύοντας την δημοκρατία και να ε, κρίνουμε σωστά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πού είναι σωστή, πού δεν είναι. Να ε, αξιολογήσουμε την ουσία της. Με αυτή την έκθεση συνδέω την ελπίδα και το αίτημα να ξεκαθαριστούν ε, ορισμένα θέματα, όπως δηλαδή ότι δεν επαρκούν οι σχέσεις όπως έχουν οριστεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και πρέπει να βελτιωθούν. Σας ευχαριστώ και εσάς. Τελευταίος είναι ο κύριος Μπρόνξ που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι σύντομος. Με ενδιέφερε πολύ η εισήγηση του κυρίου Ραγγέλ για τις άμεσες και έμεσες εκλογές για την Προεδρία ήταν πολύ εφάνταστη. Η έμεση εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν είναι δυνατή χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες. Απλώς αν εγκρίνουν τον ορισμό τον διορισμό ορισμένες πολιτικές, ό, πολιτικές ομάδες. Αλλά υπάρχει κανένα, καμία δημοσκόπηση που να δείχνει ότι το εκλογικό σώμα δέχεται να ψηφίσει τα κόμματα με βάση τον υποψήφιο που έχουν για την Κομισιόν. Νομίζω ότι το κοινό θα συνεχίσει να έχει ως βασικά κριτήρια τα εθνικά η άμεση εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν βέβαια θα σήμαινε αλλαγή των συνθήκων. Αλλά και κάτι άλλο. Υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι μεγάλο τμήμα των εκλογέων γνωρίζει αρκετά για το ρόλο του Προέδρου ή και της Κομισιόν ολόκληρης ή ακόμη και την ύπαρξη Προέδρου της Επιτροπής. για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα ψηφίσει λογικά. Εγώ φαντάζομαι ότι χωριστή άμεση εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν θα ήταν πιο εφαρμόσιμη γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ο κόσμος τι του ζητάμε να ψηφίσει. Δεύτερον, η συνθήκη της Λισαβόνας επέκτηνε τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου και εκτελεστικές και πολλοί το χαιρετίζουν αυτό, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουμε πάλι αν ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει. Όταν θα θυμάστε ο κύριος Παπαστάμκος αρρώστησε ξαφνικά στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος Σούλτς ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής και είπε ότι οι βουλευτές έχουν τόσο πολλές ψηφοφορίες που μάλλον δεν ήξεραν τι ψήφιζαν. We have to ask really why this is. Well, a lot of it's because amendments come Γιατί έρχονται οι τροπολογίες ακόμα και την τελευταία στιγμή και η βοηθή μπορεί να τις έχουν εξετάσει όλες, μπορεί και όχι, αλλά ξαφνικά την τελευταία στιγμή πάλι δύο ώρες πριν την ψηφοφορία αλλάζουν τα πάντα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και εδώ μέσα στην Επιτροπή μας έχει γίνει. Στην πρωινή μας συνεδρίαση την περασμένη Ολομέλειας. Μέχρι τις 8.30 το προηγούμενο βράδυ ελπίζαμε να κυκλοφορήσει ο κατάλογος ψηφοφορίας, δεν κυκλοφόρησε και φύγαμε. Και μετά μάθαμε ότι 12 παρατέταρτο κυκλοφόρησε. Έπρεπε λοιπόν να πάμε ταχύτατα την επόμενη μέρα να δούμε πώς θα ψηφίσουμε και ο βοηθός μου προσπαθούσε γρήγορα γρήγορα να αλλάξει τον προηγούμενο κατάλογο ψηφοφορίας. Σημείωσα όμως χωρίς να αναφέρω το όνομα του ενδιαφερόμενου κάποιον μπροστά μου που είχε προτείνει τροπολογίες και δεν τις ψήφιζε ούτε ο ίδιος. Αναρωτιέμαι γιατί, μάλλον δεν τις αναγνώριζε. Ας μην επαναλάβω τις απόψεις μου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις έχω πει πολλές φορές, αλλά η ψηφοφορία σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο πρέπει να γίνεται μετά από επαρκή πληροφόρηση. Τέτοιου είδους διαδικασίες δεν είναι λογικές. Ξέρουμε ότι οι αρχηγοί των κομμάτων δείχνουν στους συναδέλφους τους πώς να ψηφίσουν, αλλά αν δεν έχουν αποφασίσει μόνοι τους, τότε πώς θα δεχτούν απλώς τι τους λένε. Εγώ είμαι στην αξιοζήλευτη θέση να μην υπόκειμαι σε τέτοιες πιέσεις και κοιτάζω μόνο με τους βοηθούς μου να δω κάθε φορά πώς θα ψηφίσω. Αλλά βέβαια δεν μπορεί κανείς να είναι παντού ταυτόχρονα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις βιαστικές συνεννοήσεις με τους βοηθούς που χρειάζεται καμιά φορά να ικανοποιήσουν δύο αντίθετες απόψεις. Ας μην συνεχίσω. Καλώς, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Ή αν συνάδελφος Ραντζέλ θέλει να αντιδράσει στα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Ραντζέλ. Ε, ε, θα απαντήσω πολύ σύντομα. E Υπάρχει μια ιδέα που σημαίνει ότι Άντριου Ντόφ και ο κύριος Μορέιρα ε, μοιράζονται. Δηλαδή ποια είναι η ακριβή κάλυψη που θα έχει αυτή η έκθεση. Ποια είναι τα πλαίσια στα οποία Νομίζω ότι ο συνάδελφό μα ο κύριος Σόλτς έχει απόλυτο δίκιο στα όσα μα είπε. Αν η δουλειά μα εδώ είναι να κάνουμε Ετοιμάσουμε άλλη μία διοικητική φύσεω έκθεση στην Επιτροπή Στεματικών Υποθέσεων, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι αν είναι απλό ζήτημα διοικητικών εκθέσεων, τέτοιων απλών εκθέσεων, αυτό μπορεί να γίνει και από κάποιο μέλος της διοίκησης και όχι από κάποιον πολιτικό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι πολιτική φύσεως έκθεση. Αν δούμε τις εφαρμοστικές πράξεις, τις κατεξουσιοδότησης πράξεις, το ρόλο του κοινοβουλίου, του Ελέγχου κλπ. Αυτά θα έχουν πολιτικές συνέπειες και γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε στις πολιτικές συνέπειες εξετάζοντάς σωστά από πολιτική σκοπιά. Και αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι κάτι αποκλειστικά διοικητικό. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να αλλάζουμε ένα σύστημα. Και αυτή η αλλαγή θα έχει πολιτικές συνέπειες. Δεν ζητείτε να προβούμε σε μία αποτίμηση της συνθήκης της Αβώνας, αυτό που αναφέρεται στο τίτλο και μόνο, εγώ δεν θα παραιτηθώ του δικαιώματος να αξιολογήσω τα πράγματα συνταγματικά και πολιτικά και να εξετάσω τα αποτελέσματα της συνθήκης της Αβώνας από αυτή την οπτική γωνία. Και μάλιστα διότι αυτό περιμένει ο κόσμος από εμά. Δεν περιμένουν από εμά να αναφερθούμε στις διοικητικές αλλαγές, να πούμε χ, ψ, ω, αλλαγή, άρα πρέπει να κάνουμε χ, ψ, ω, αλλαγή και εμείς είναι σαφές ότι και αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει, όμως είναι πολύ πιο σημαντικό για μας να προσεγγίσουμε το ζήτημα από μια πιο μακροσκοπική προσέγγιση και ε, να μπορέσουμε να κάνουμε ε, από το γράφημα στο οποίο θα καταλήξουμε να κάνουμε μια επέκταση του γραφήματος, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μέσω μιας ε, παρεκφολής. νομίζω ότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή βλέπουμε να υπάρχει μια τριάδα που δημιουργείται. Πολλαπλές κυβερνήσεις από τη μια πλευρά, ε, μετά σχέσεις με το Συμβούλιο και μετά σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν περιοριστούμε και μπούμε στις λεπτομέρειες, θα χάσουμε ευρύτερα ζητήματα. Θα έχουμε μια έκθεση για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, θα έχουμε μια άλλη για άλλες λεπτομέρειε και μια διοικητική φύσεως έκθεση, η οποία απλώς θα προέβαινε σε μια αποτίμηση των αλλαγών ε, που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνα αφορά το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα χρειάζεται ευρύτερη προσέγγιση, γενικότερη εικόνα. Αυτό δεν είναι κάτι που υπονομεύει τα όσα είπε και ο Σβιτάλ Μορέρα. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κ. Μορέιρα έχει δίκιο, απόλυτο, που είπε ότι νομοθετικά ζητήματα πρέπει να διαχωριστούν από διοικητικά και τεχνικής φύσης ζητήματα. Όμως, παρόλα αυτά χρειάζεται γενικότερη προσέγγιση. Ολιστική προσέγγιση. Γι' αυτό ακολούθησα αυτή την προσέγγιση. Αν ακολουθήσουμε μια πιο λεπτομερή προσέγγιση θα είναι ασφαλμένο και καλύπτει μόνο μια σκοπιά. Απαντώντας τον κύριο Νταφ, συμφωνούμε ουσιαστικά όσον αφορά τι κατεξισοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις. Συμφωνώ βασικά με όλα όσα υπόθηκαν. Όταν αναφέρθηκα στη θεωρία της του ουσιαστικού χαρακτήρα των πραγμάτων, το ανέφερα διότι η εάν η διαμόρφωση πολιτικής περνάει μέσα από της πράξης πρέπει να γίνεται για κάποιο λόγο. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα θέματα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και γι' αυτό ανέφερα και το πολιτικό ζήτημα και ότι χρειάζεται κοινοβουλευτική διακυβέρνηση. Αν το κοινοβούλιο ε, θεσπίζει επί λεπτομεριών νομοθεσία, τότε θα γίνεται διοικητική δουλειά και όχι πολιτική νομοθετική. Γι' αυτό χρειάζεται διαχωρισμός των καθηκόντων αυτών. Και πρέπει να καταλάβουμε και ποιες είναι οι συνέπειες των αλλαγών. Και στην ομάδα το συζητήσαμε το θέμα. Κάτι που ανέφερε ο κύριος Ντόφ και κάτι άλλο που ανέφερε ο κύριος Βιτάλ Μορέιρα που αναφέρθηκαν σε πολιτικά ζητήματα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου δεν ξέρω ποιος να το αναφέρει αυτό το θέμα. Υπάρχει σύγχυση εξουσιών. Χρειάζεται αλλαγή. Στην αρχική μου παρουσίαση αναφέρθηκα στο Ενωμένο Βασίλειο που σε κάποια φάση ο βασιλιάς ήταν στο κοινοβούλιο σε κάποια φάση ιστορίας και τώρα θα έχουμε ένα κοινοβούλιο που θα βασιλεύει το ΣΥΠΗΝ περίεργο μόρφωμα αυτό Πιστεύω όμως ότι είναι χρήσιμη η αλλαγή, είναι χρήσιμες οι αλλαγές που έγιναν. Συχνά όμως όταν γίνονται χρήσιμα πράγματα επηρεάζονται οι αρχές που κρύβονται πίσω από αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να θυμόμαστε τις αρχές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Φερρυπίν να παρίσταται σε σημαντικές εκδηλώσεις εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να είναι νομοθετικός φορέας πραγματικά με σημαντικό ρολό όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να κάνει τη δουλειά που τον ετέθη. Είναι σημαντικό. Έγιναν αλλαγές, αυτό πρέπει να δούμε, αλλά δεν είναι αρκετέ ακόμα. Αυτό που αναφέρθηκε μετά, η νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα, τα ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι περισσότεροι θα έλεγαν ότι το θέμα του νόμου για τα πολιτικά κόμματα δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε θετική λύση του προβλήματος. Θα δούμε τα αποτελέσματα στις επικείμενες ε, εκλογές. Δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά, νομίζω θα αποτύχουμε. Στο ΕΛΚ και εγώ και συνάδελφοι υποβάλαμε αρκετές τροπολογίες για να αλλάξουμε την κατάσταση. Το ελικό αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι είναι καλό για τα πολιτικά κόμματα. Αντίθετα με την προηγούμενη ερώτηση και το προηγούμενο ζήτημα, δεν ξέρω κατά πόσο η εξέλιξη θα είναι θετική για το Κοινοβούλιο μακροπρόθεσμα στο συγκεκριμένο θέμα αν δούμε τι αντίκτυπο θα έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ εστιάζεται και η έκθεση. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κατά πόσο οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επηρεαστούν αρνητικά. Αυτό που δημιουργούμε είναι μια υποδομή εντός του συνταγματικού μας μοντέλου. Και πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς πού εντάσσονται όλα τα στοιχεία στην υποδομή Αλλιώς θα χαθεί κάθε έλεγχο. Απαντώντας τον κύριο Σόλτς, συμφωνώ ότι πρέπει να εντοπιστούν πολιτικά και συνταγματικά ζητήματα πριν προχωρήσουμε. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Μπρόντς, ήσασταν μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, κύριε Μπρόντς. Α, ναι, το βλέπει κανείς αυτό. Διότι αν υπήρξατε μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου θα καταλαβούσατε πώς λειτουργεί. Ακούμε διάφορε και σχόλια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσεί θα έπρεπε να διαμαρτύρεστε για τον τρόπο λειτουργία του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Έλεγα στον συνάδελφό σα, τον κύριο Φόξ, ότι ίσω θα έπρεπε να πάτε στο Westminster, να πάτε, να πηγαίνετε αρέα και που για να δείτε πώ λειτουργεί. Τι θα βλέπατε εκεί. πραγματικά, αν θεωρείτε ότι αντικατοπτήσετε πραγματικά η δημοκρατία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ελάτε, πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται εκεί και μετά να έρθετε εδώ να μας επικρίνετε. Ο κύριος Μορέρα αναφέρθηκε ότι υποστηρίζει την κοινοβουλευτική προσέγγιση. Το ξέρω, το ξέρω καλά, αλλά υπάρχει κάτι που είναι ξεκάθαρο. Στο μοντέλο διακυβέρνησης για μεγάλες χώρες και μεγάλες περιφέρειες βλέπουμε ότι τα περισσότερα είναι προεδρικά και σχεδόν όλα είναι προεδρική φύσεω και δεν τυχαίο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ ποικιλόμορφο. Και ίσως να λειτουργεί καλύτερα με βάση το κοινοβουλευτικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο λόγω ε, μεγέθους. Αλλά λόγω ποικιλόμορφίας των περιφερειών που εκπροσωπούνται, ίσως να μην λειτουργήσει καλά. Να λειτουργεί καλύτερα το προεδρικό σε άλλε περιοχέ, Ηνωμένε Πολιτείε, Πολιτείες, Ινδία κλπ. βλέπουμε ότι λειτουργεί καλύτερα το προεδρικό. Σε μεγάλε περιοχέ, σε μεγάλε χώρε λειτουργεί καλύτερα το προεδρικό μοντέλο. Αυτή είναι η τάση. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν την περιγράψω και στην έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου. Όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου τη Κομισιόν, ο κύριο Μπροντ, λέει κάτι που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον. Λέει, εάν ο πρόεδρο δεν εκλέγεται άμεσα, αλλά έμεσα δεν θα ξέρεις ακριβώς ποιος είναι, ποιοι είναι για, για πρόεδρο και το εκλογικό σώμα δεν γνωρίζει κάτι, σύμφωνα με τον κύριο Μπρόντς. Εμείς πρέπει να κάνουμε επιλογή. Να πούμε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει. Πρέπει να αποφασίσουμε, δίνουμε στους πολίτες το δικαίωμα να επηρεάσουν την εκλογή του Προέδρου μέσω του Κοινοβουλίου ή μέσω προεδρικών εκλογών με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες δικαίωμα λόγου όσον αφορά τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαφορετικά επιτρέπουμε να εκλέγεται ο Πρόεδρος άνευ Αν έχουμε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξάρτητα αν κάποιος ξέρει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και ποιος είναι, παρόλα αυτά θα υπάρχει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσως τεχνοκράτης. Εάν εμπλακούν μέσω εκλογών οι πολίτες, ίσως αποκτήσουμε επαφή με τους πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συχνά οι πολίτε δεν γνωρίζουν. Αν υπήρχαν άμεσε εκλογέ, θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται και οι πολίτε στι ΗΠΑ. Που είναι ενωμένε πολιτείε και ίσω θα είναι καλό μοντέλο και για μα, για το Σύνταγμά μα. Πολλοί δεν ψηφίζουν τι προεδρικέ εκλογέ. Δεν του ενδιαφέρουν οι προεδρικέ εκλογέ και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πιο ομοιογενεί από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο, ο, πρόεδρος της, ε, των Ηνωμένων Πολιτείων στερείται νομιμότητας. Όχι. Ο πρόεδρος την χάνει ευρείας υποστήριξης των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε είναι από τη Νότια Καρολίνα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Ουάσιγκτον, την Καλιφόρνια, δεν τους νοιάζει. Αυτό που τους νοιάζει είναι τι κάνει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό γίνεται στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν και παραπάνω λόγοι παρόμοιες προσέγγισης εδώ από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Λέγεται ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για εθνικά ζητήματα. Ναι, πράγματι. Αλλά αν συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι έτσι πετυχαίνουμε καλύτερη δημοκρατία. Λέω λοιπόν ότι αν έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν υπάρχει, εγώ προτιμώ να είναι δημοκρατικά εκλεγμένος παρά το αντίθετο. Πώς θα συμβεί αυτό. Αυτό εξαρτάται από τους πολίτες. Ξέρω τι θα ήθελαν κάποιοι. Να απαλλαγούν από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα θέλαν. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Θα έχουμε πρόεδρο. Πώ θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αυτή είναι η απάντηση προ τον κύριο Μπρόν. Δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να το απαντήσω. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι απάντησα αρκετά. Πρόεδρε, θα πάω σπίτι μου, θα σκεφτώ αυτά που ακούστηκαν, θα προσπαθήσω να ετοιμάσω κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα είναι αρκετά δύσκολη η δουλειά όπως και το χρονοδιάγραμμα που είναι περιοριστικό αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους και να ολοκληρώσουμε στη θητεία μας αυτό, αυτή τη σημαντική έκθεση χρειάζεται να έχουμε ρυθμό εντατικό. Προτείνω λοιπόν να γίνουν τα εξή. 17 Δεκεμβρίου του 2013 φέτος υποβολή του σχεδίου γνωμοδοτήσεως κύριε Ραντζέλ. Ακρόαση δημόσια 20 Ιανουαρίου 23 Ιανουαρίου του επομένου έτους προθεσμία για κατα... υποβολή τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Ολομέλεια Μάρτιος του 2014. Βλέπω να γνέφεται καταφατικά, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αυτό απεφασίστη. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το σημείο που ο κύριος Μέσσερ Σμιτ ε, θα είχε θέσει, γιατί είναι... Γιατί να τα αναβάλουμε για αύριο. Λίγο λεπτό λίγα λεπτά για να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είμαι εισηγητή, που είναι το σημείο 7 τη ημερήσια διατάξη τη αρχική, δηλαδή είναι η ερμηνεία του άρθρου 202, παράγραφο 5 του κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τι αποστολέ συλλογή πληροφοριών. Ασχολούμεθα με αυτό. Εγώ επελήφθην ε, με την προετοιμασία μια γραπτή γνωμοδοτήσεω που μπορούμε, αν θέλετε, να ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Και έχω κάτι σχετικά απλό Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το ιστορικό. Η Επιτροπή των Αναφοράν μας ζήτησε ε, μία ερμηνεία του άρθρου 202 όσον αφορά τι συγγύες που πρέπει να κάνει, τι εκθέσει που ετοιμάζει η Επιτροπή μετά από τι αποστολέ που κάνει όσον αφορά την επαλήθευση επιτόπου. Να πηγαίνει σε μία άλλη χώρα, σε μία άλλη περιφέρεια για να κάνει μία επαλήθευση μια καταστάσεω, να συλλέξει στοιχεία για να τοποθετηθεί και να καταλήξει συμπεριέσματα κατόπιν μια υποβολή αναφορά από πολίτε. Λοιπόν, στην παράγραφο 5 του άρθρου 202 αναφέρει τα εξή και διαβάζω για τους σκοπούς εξέτασης αυτών των αναφορών και την επιβέωση των στοιχείων ή προς την προσπάθεια εξέβασης λύσεων, η Επιτροπή μπορεί να οργανώνει αποστολές ενημέρωσης στο κράτος μέλος ή στην περιφέρεια όπου αναφέρονται στην ε, αναφορά. Οι εκθέσεις για τις αποστολές ε, συντάσσονται από τους συμμετέχοντες. Αυτές διαβιβάζονται στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου μετά από την έγκριση της Επιτροπής. Γιατί η Επιτροπή των Αναφορών μας ζητά αυτή τη γνωμοδότηση, μας ζητά να δώσουμε ερμηνεία, διότι μετά από μία αποστολή στη Γαλλικία, οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία που πήγε εκεί, δεν συμφώνησαν όσον αφορά τη σύνταξη της εκθέσεώς τους. Και ούτε η Επιτροπή στο σύνολό της κατάφερε να εγκρίνει. Δεν ήξερε ποιον κανόνα να εφαρμόσει. Η πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει την εφαρμογή του άρθρου 52, αλλά το άρθρο 52 αναφέρεται σε άλλα θέματα αναφέρεται στις ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ μιλάμε αντιθέτως για μια φάση μιας διαδικασίας που είναι τυπική διαδικασία όσον αφορά την Επιτροπή των Αναφορών που ολοκληρώνεται με μια έκθεση που αποστέλλεται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφέρεται στο 202 ρητά ότι η έκθεση όσον αφορά την αποστολή συντάσσεται από τους συμμετέχοντες δεν λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία και εδώ ακολουθώ τη γνωμοδότηση που δόθηκε από την νομική υπηρεσία φαίνεται ότι αυτή η έκθεση όσον αφορά τα όσα συνέβησαν και στην αξιολόγηση των όσων έγιναν στην αποστολή θα πρέπει να είναι αντικείμενο συνένεση. Μάλλον λόγια πρέπει να εγκρίνεται από όλα τα μέλη τη αντιπροσωπεία. Σαφώ, αν αυτό δεν συμβεί, ο καθένα καταγράφει τα στοιχεία όπως τα είδη τα πράγματα και όπως τα αξιολογεί. Όλα αυτά γράφονται και συνένεση αφορά μόνο ότι καταγράφονται οι διάφορες απόψεις όσον αφορά την αξιολόγηση και τα στοιχεία. Όμως το άρθρο συνεχίζει και λέει, το άρθρο 202 και λέει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει. Άρα πρέπει να γίνει ψήφος έγκρισης που δεν μπορεί παρά να είναι ομόφωνη. Και ε, μάλλον να γίνεται μια ψηφοφορία μοναδική και να επικρατήσει η πλειοψηφία. Εκτός εάν η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου λέει αν θεωρεί ο Πρόεδρος ότι επιτρέπονται τροπολογίες. το τέλος όμως θα γίνει μια ψηφοφορία και αν δεν γίνει η ψηφοφορία, δεν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, καμία έκθεση δεν θα υποβληθεί από την Επιτροπή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και όλα λήγουν. Εδώ σας δείχνω γραπτά την ε, γνωμοδότηση στο φάκελό σας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε εκτός από κάτι. Στο τελευταίο τμήμα της γνωμοδοτήσεως λέει ότι, πρέπει να βρω που το λέει, ότι οι αποστολές ενημέρωσης και τα πρακτικά, διαβάζω εδώ που είναι, αν θέλετε μιλάτε πάνω σε αυτό. Οι αποστολέ αυτές και τα πρακτικά αυτά της επίσκεψης έχουν σαν μόνο στόχο να δώσουν στην Επιτροπή αναφορών σε αυτή την περίπτωση τις αναγκαίες πληροφορίες ούτως ώστε να εξεταστεί αναφορά. Γι' αυτό τα πρακτικά συντάσσονται από, την, από τους συμμετέχοντες που θα πρέπει να προσπαθήσουν να καταλήξουν στη συνένεση. Ελείψει τέτοια συνενέσεως η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις διάφορες διαπιστώσεις και τις εκτιμήσεις ε, τις αποκλίνουσες. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή των Αναφορών προς έγκριση μέσω μιας ψηφοφορίας εκτός και αν ο πρόεδρος δηλώνει, όποτε αυτό ενδείκνυται, ότι η κατάθεση τροπολογιών μπορεί να γίνει για κάποια τμήματα της εκθέσεως. Το άρθρο 52 δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις εκθέσεις ούτε άμεσα ούτε έμεσα ελήψη, εδώ, το κείμενο που έχετε εσείς στο φάκελό σας λέει, ελήψη συνένεση μεταξύ των συμμετέχων ή εγκρίση από την Επιτροπή, εκθέσεις δεν θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις εκεί που λέει ελήψη συνενέσεως μεταξύ των συμμετέχοντων ή όχι. Μπορεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ε, συμμετοχόντων. που λέει ελλείψη συνενέσεω τι γίνεται. Εγώ θα το διάγραφα αυτό που τι γίνεται ελλείψη συνενέσεω. Και το τελικό τμήμα θα μείνει ω έχει. Ελλείψη εγκρίσεω από πλευρά τη επιτροπή καμία έκθεση δεν διαβιβάζεται στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Να παραμείνει αυτό. Αν θέλετε να μιλήσετε όσον αφορά αυτή την άποψη, που εγώ προτείνω να τη διαβιβάσουμε όπως σας τη διάβασα, γραπτός με τη διόρθωση, και ψηφίζουμε αύριο το πρωί, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος. Βλέπω κάποιο χέρι να έχει σηκωθεί. Θέλετε το λόγο. Ορίστε. Ε, κυρία Πέτροβιτς, ζητήσατε να μιλήσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Από την προηγούμενη συζήτηση στην προηγούμενη συζήτηση είχαμε ακρηγορήσει. Θέλω απλώς τώρα να πω ότι ως σκιώδης εγκρίνω την γνωμοδότησή σας για την ερμηνεία του άρθρου 22. Ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης δεν απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και δεν μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες γιατί αφορά γεγονότα Γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως τη λογική που εκφράζεται στην επεξηγηματική έκθεση του γράμματός σας κύριε Πρόεδρε. Και όλα αυτά μπορούν να διευκολυνθούν όταν δίνεται δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν και διαφωνούσες απόψεις εφόσον βασίζονται σε διαφορετικές διαπιστώσεις. Αυτό θα διασφάλιζε ότι όλοι θα γνωρίζουν όλες τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που έχουν γίνει και άρα θα συμφωνούσε πλήρως με τη λογική του κανονα 2.2 για την μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Αναλογικά, το περιεχόμενο της έκθεσης δεν μπορεί να ψηφιστεί μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας γιατί τότε η ΑΝΑΦ δεν θα μπορούσε να έχει όλα τα στοιχεία. Η επεξηγηματική σας έκθεση κύριε Πρόεδρε είναι εξαιρετική εξήγηση των λόγων για την ερμηνεία αυτή και γενικά θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ο συνάδελφος Μπρόν συζήτησε το λόγο. Βρήκα την απάντηση στο ερώτημά μου, οπότε δεν θέλω να μιλήσω. Καλώ, δεν βλέπω άλλους να θέλω να μιλήσουν. Θα ψηφίσουμε αύριο στην Ολομέλεια της Επιτροπής και εδώ Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση απογευματινή. Υπενθυμίζω δύο πράγματα σημαντικά. Πρώτον, αύριο το πρωί θα διεξαχθεί η συνεδρίαση των συντονιστών 9 και στις 9 και 50 θα ξεκινήσει η Επιτροπή της Εργασίας. Δεύτερον, το απόγευμα θα υπάρξει αυτό το σεμινάριο, ιδιαίτερα σημαντικό σεμινάριο, όπου εκεί θα διεξαχθεί διάλογος η προσαξιολόγηση από κοινού με την κοινωνία των πολιτών πιο συγκεκριμένα με τους φιλοσόφους, θρησκευτικού ηγέτες και με τους κοσμικούς εκπροσώπους την κατάσταση ε, που, διαμορφώνεται πριν από τις εκλογές. Πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλλει ούτω ώστε να έχουμε επιτυχία όσον αφορά τη συμμετοχή στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.